Ε, euh, Ωραία λοιπόν, θα αρχίσουμε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχουμε πολύ βαρύ πρόγραμμα σήμερα. Γι' αυτό θα είμαι σύντομη και μετά θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας που τους ευχαριστώ για την προσέλευσή τους στην ακρόαση αυτήν. Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης έχει ως στόχο, όπως γνωρίζετε, να χορηγεί βοήθεια επιγόντως για να ανταποκριθεί σε ανάγκες και να προστατευτούν ζωές. Η δυνατότητα των ανθρωπιστικών παραγόντων για χορήγηση βοήθειας ουδέτερα αντικειμενικά και ανεξάρτητα αμφισβητείται όλο και περισσότερο από πολιτικές, στρατιωτικές και ασφαλιστικές σκέψεις οι εντολές των στρατιωτικών και ανθρωπιστικών αποστολών σε περιφέρειες που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή σειράξεις πρέπει να είναι σαφείς. <clears throat> Τα μέσα και οι στρατιωτικές δυνατότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και σύμφωνα με τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών. Παρόλα αυτά υπάρχουν καταστάσεις όπου μια στρατιωτική παρέμβαση θα μπορούσε να βοηθήσει την ανθρωπιστική όπως στην Αϊτή. Η πρόσβαση στους ε, πληγέντες πληθυσμούς είναι όλο και πιο δύσκολη και η ασφάλεια των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν είναι εγγυημένη. Η ανθρωπιστική διάσταση στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και θα έπρεπε να περνάει από μια ευαισθητοποίηση του κόσμου προς τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει έκθεση πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Συνένεση για τα ανθρωπιστικά στο Συμβούλιο και την Κομισιόν όπου ζητήσαμε να υπάρξουν σαφείς κανόνες για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών για την Εξωτερική Δράση και της Κομισιόν για τη διαχείριση μεγάλων κρίσεων. Η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει δράσεις ευαισθητοποίησης για την ανθρωπιστική δραστηριότητα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάλογο μεταξύ στρατιωτικών και ανθρωπιστικών παραγόντων που είναι τελείως απαραίτητος για να προωθηθεί μια αμοιβαία κατανόηση. Χωρίσαμε σε τρία μέρη την ακρόαση αυτή. Κάθε πάνελ θα ακολουθείται από ερωταπαντήσεις. Για το πρώτο βάλαμε ως τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση και Διαχείριση Κρίσεων Μήπως υπάρχει κίνδυνος πολιτικοποίησης ή στρατιωτικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Χρόνος 9 και 20 με 10 και 40, μία ώρα και 20 λοιπόν. Και στο πρώτο αυτό πάλι θα μιλήσουν τέσσερις. Πρώτον ο κύριος Ρος Μάουντεν, Γενικός Διευθυντής της Δάρας, που θα μας κάνει μια γενική εισήγηση για την πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μετά η κυρία Εστέρα Σιν Μαρτίνες, εκπρόσωπο της Care International που θα μας παρουσιάσει την άποψη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και μετά ο κύριος Πέτερ Τσάγκλ, Γενικός Διευθυντής της ΕΚΟ. Τελευταία δε, ο κύριος Μιότσο, που είναι Διευθυντής της Υπηρεσίας για την εξωτερική, χορήγηση της εξωτερικής βοήθειας. Ο κάθε ομιλητής και ομιλήτρια πρέπει να γνωρίζει ότι έχει μετρημένο χρόνο ο καθένας έχει 8 λεπτά. Παρακαλώ να σεβαστείτε αυστηρά τον χρόνο αυτόν, ώστε να μπορέσουν όλοι και όλες να συμμετάσχουν όπως πρέπει. Ο κύριος Ρος Μάουντεν λοιπόν αρχίζει. Σας κατευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο που ζητήσατε αλλά θα είναι δύσκολο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να προσέλθω εδώ. Βλέπω διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ μέσα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει, ιδίως στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για την <clears throat> ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς δεχόμαστε την έκθεση για τα συμπεράσματα του, ε, της Ευρωπαϊκής Συνένεσης που συμφωνούν σε πολλά με τα δικά μας. Η έκθεση ταυτίζει σωστά την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση και γνώση των ανθρωπιστικών αρχών μεταξύ κυβερνήσεων και υπηρεσιών όπως την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία και συμφωνούν και με την αναθεώρηση που έκανε πρόσφατα η Βρετανική κυβέρνηση για την ανθρωπιστική της ανταπόκριση. Γιατί είναι σημαντικό το θερινό μας θέμα. Η οργάνωσή μου η Δάρα γράφει κάθε χρόνο μία έκθεση για την ανθρωπιστική δράση και το κατά πόσον γίνονται σεβαστές οι σωστές αρχές ανθρωπιστικής δωρεάς ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες και μόνον σε αυτές και μάλιστα ακολουθεί τις βασικές αρχές ουδετερότητας που ανέφερε προηγουμένως και η Πρόεδρος. Τα περσινά μας συμπεράσματα, το 2010 δηλαδή, ήταν ότι η πολιτικοποίηση και εκμετάλλευση της βοήθειας είναι πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται. 10 από τις 14 χώρες που μελετήσαμε έδειξαν σημεία τάσης πολιτικοποίησης είτε από τις κυβερνήσεις που κάνουν τις δωρεάς είτε από άλλους παράγοντες. Και αυτά προκύπτουν από αναθεωρήσεις που έκαναν οι ίδιες οι χώρες στο διαδίκτυο καθώς και μη κυβερνητικοί παράγοντες. Η κυριότερη ανησυχία μας είναι ότι η στρατιωτικοποίηση της βοήθειας ιδίως σε περίπτωση σειράξεων μπορεί να έχει μεγάλες αρνητικές, σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την προστασία των αμάχων. Αυτό το μείγμα στο Αφγανιστάν έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο τις ζωές των ε, εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Μερικές κυβερνήσεις έχουν πάρει σαφή θέση για την προστασία του ανθρωπιστικού χώρου και την προώθηση των ανθρωπιστικών αρχών, μεταξύ αυτών και το Κοινοβούλιο με τις εκθέσεις του, καθώς και η κυβέρνηση του ΙΤΑΒ. Για την ΕΕ θα ήθελα να σας σχολιάσω τι έκανε η ΕΚΟ που μέχρι στιγμής έχει σεβαστεί τις βασικές ανθρωπιστικές αρχές της χορήγησης βοήθειας με βάση τις ανάγκες και με ουδετερότητα, ακαιρεότητα και ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας χωριστά από οποιοδήποτε άλλο στόχο. Η ΕΚΟ δεν είναι ο μόνος παράγοντας που τα εφαρμόζει αυτά. Μερικές όμως κυβερνητικές υπηρεσίες υπονομεύουν τις αρχές αυτές και δεν χρησιμοποιούν σωστά τις ανθρωπιστικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οφείλεται σε έλλειψη γνώσης ή κατανόησης του ποια είναι η ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής βοηθείας και τι ρόλο ακριβώς παίζει και γιατί, γίνεται, γιατί υπάρχουν τα συμπεράσματα της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης που μιλάν για την ανάγκη εφαρμογής αυτών των αρχών. Το συγκεκριμένο θέμα του συνδυασμού πολιτικής και στρατιωτικής βοήθειας είναι κάτι που δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αποκλείεται, ούτε είναι ασύμβατα αυτά τα δύο, εξαρτάται από τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, είναι βασικό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός, διάκριση μεταξύ στρατιωτικών και ανθρωπιστικών παραγόντων και ότι οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών πόρων για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν μη στρατιωτικά μέσα στη διάθεσή μας και πάντοτε υπό πολιτική και όχι στρατιωτική ηγεσία. Αυτό ίσως θα πρέπει και να το τονίσουμε. Η έλλειψη διαχωρισμού μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού σκέλους μπορεί να έχει πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη διασφάλιση της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο Αφγανιστάν έχουν σημειωθεί περισσότερες παραβάσεις και παραβιάσεις. Μπορεί να υπάρχουν εθνικές στρατιωτικές υπηρεσίες που δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα εδώ των χωρών των ίδιων όπου σημειώνεται η κρίση ή συγκεκριμένες μεμονωμένες κυβερνήσεις με ή χωρίς εντολή του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι ίδιες οι δυνάμεις ασφαλείας του ΟΗΕ που μπορούν να αναλάβουν το στρατιωτικό σκέλος. Οι κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο και οι πιο ενημερωμένες και σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατιωτική και πολιτική βοήθεια ε, αποτελούν ένα πλαίσιο για την... που μπορεί να μας οδηγήσει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα καταχρήσεων. Ένα είναι η αντιμετώπιση θεομηνιών όπου εθνικοί πόροι μπορεί όπως το Πακιστάν να χρησιμοποιηθούν με πολύ θετικά αποτελέσματα αλλά αυτό εξαρτάται από τους πόρους ακριβώς που διαθέτει κάθε χώρα. Υπάρχουν και άλλες στηρικτικές δομές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπως στην IT ή στην αντιμετώπιση του τσουναμίου. Οι σειράξει είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολλές φορές υπάρχει δύναμη με εντολή του ΟΗΕ, σαφή εντολή, <coughs> για τη διασφάλιση της προστασίας των αμάχων, όπως στη δημοκρατία του Κονγκό, τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και πρέπει και αυτές οι δυνάμεις να γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τους διότι η προστασία των προσώπων είναι ο κανονικός ρόλος του στρατού, των στρατιωτικών δυνάμεων και όχι η χορήγηση ανθρωπιστικής βοηθείας. Για τις σειράξεις μπορεί ένα από τα δύο μέρη, είτε η κυβέρνηση είτε οι εξεγερμένοι, να μη σέβονται τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση της ανθρωπιστικής βοηθείας και είναι από τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουμε για να διασφαλιστεί, που, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντοτε, η ουδετερότητα της χορήγησης βοήθειας παράδειγμα το Αφγανιστάν. Για τη χορήγηση αυτής της ανθρωπιστικής βοηθείας το βασικό θέμα είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι ανάγκες του πληθυσμού που θέλουμε να προστατεύσουμε με στόχο πάντοτε την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς μας που δεν πρέπει να βασίζεται στο τι έχουμε να προσφέρουμε αλλά στις ανάγκες τους. Συνήθως ο ΙΕΟ, ο Ερυθρός Σταυρός, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν τις δυνατότητες που πρέπει και τους πόρους για να αναλάβουν τη χορήγηση της βοηθείας. Αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο στρατός. Εδώ υπάρχει η ανησυχία του πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον για τη Λιβύη ας πούμε. Εκεί μπορεί να υπάρξει ανάμιξη του πολιτικού με τον ανθρωπιστικό στόχο. Αλλά πρέπει ο καθένας να γνωρίζει σαφώς τα όρια του. Σε μερικές κρίσεις που μελετήσαμε υπήρξαν κυβερνήσεις που ρητά ζήτησαν από, το από τις στρατιωτικές τους δυνάμεις να κάνουν και ανθρωπιστικό έργο ή έργο σταθεροποίησης και αντιμετώπισης ε, εξεγέρσεων. Αυτά δεν είναι ανθρωπιστική στόχη βέβαια. Υπάρχει και μια εκμετάλλευση που μπορεί να γίνει των ανθρωπιστικών στόχων όπως αν οι δωρητές δώσουν την προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη και όχι στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης όπως στην Κολομβία και τη Σομαλία. Η χρηματοδότηση και στήριξη κυβερνήσεων θα πρέπει να έχει υπεύθυνου από τις κυβερνήσεις αυτές όπως στη Ζιμπάμπουε αλλά δεν είναι δυνατόν να αγοράσει κανείς και την καλή θέληση για τις χώρες που χορηγούν την βοήθεια είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με τις ειδικευμένε ανθρωπιστικές οργανώσεις για να αποφευθεί ο κίνδυνος άθελης, αθέλητης ε, χειροτέρευσης της κρίσης. Δεν έχω χρόνο να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί και μη κυβερνητικοί και κυβερνητικοί παράγοντες μπορούν να πολιτικοποιήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Και τελειώνω λέγοντας ότι η υποστήριξη της βοήθειας με ανθρωπιστικές αρχές είναι κάτι το σωτικό όχι μόνο λόγω των αρχών, αλλά και για πρακτικούς λόγους. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών μελών πρέπει να είναι να ζητούν πάντοτε την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ανθρωπιστική βοήθεια και να διασφαλίζουν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες και οι διπλωματικές προσπάθειες θα υποστηρίζουν τις καθαρά ανθρωπιστικές και τελικά η αποτελεσματικότητα είναι το ουσιαστικότερο κριτήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάουντιν. Η κυρία Μαρτίνες έχει το λόγο τώρα. Um, thank you very much, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Στρίφλερ και ευχαριστώ την Επιτροπή ΔΕΒΕ που οργάνωσε αυτή την ακρόαση σήμερα για να ορίσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Και τις υπόδομες ονομάζομαι Στρέλα Μαρτίνες ε, Εργάζομαι για μία μη κυβερνητική οργάνωση που ε, εργάζεται σε 87 χώρες με ανθρωπιστική, για ανθρωπιστική βοήθεια και για βελτίωση της ζωής των φτωχότερων, ιδιαίτερα των ε, γυναικών και των παιδιών. Είμαστε στο Voice και σε διάφορα ε, δίκτυα δίκτυα τα οποία ε, διασυνδέονται και με τα ΜΜΕ. Όπως ξέρετε, η πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας μας απασχολεί ιδιαίτερα. Όχι επειδή δεν μας αρέσει να πολιτικοποιείται, αλλά για πρακτικούς λόγους. Όπως είπε ο κ. Μάουντεν, έχει να κάνει με την ασφάλεια του προσωπικού και των δικαιούχων που αυτοί αντιμετωπίζουν ε, άμεσα τις απόρριες της πολιτικοποίησης, αυτής της συνέπειες της ε, πολιτικοποίησης αυτής, όπως είδαμε πρόσφατα στο Αφγανιστάν. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ακριβώς επειδή διαφέρουμε από άλλους φορείς ιδιαίτερα στρατιωτικούς. Γι' αυτό η διαχείριση αυτών των, αυτής της σχέσης θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση και να μπορούμε να βοηθούμε αυτούς που χρειάζονται τη βοήθεια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με προσοχή. Νομίζουμε ότι ε, ο, αυτή η κατάσταση τρόμου και δέους οδήγησε σε μεγάλες δυσκολίες και ως προς τη χορήγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος και οργανώσαμε όπως την ΚΕΡ και άλλων που δρούν επιτοπίως. Ως προς την συνολική αυτή προσέγγιση είναι ένα βασικό δόγμα, αποτελεί βασικό δόγμα του ΝΑΤΟ αλλά και μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η συνεκτική αυτή προσέγγιση αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη κατά πιο ε, συνεκτικό τρόπο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Φολκ όρισε ότι οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να δώσουν ολοκληρωτικές απαντήσεις. Χρειάζεται η υποστήριξη διεθνών οργανώσεων και μη κυβερνητικών έτσι ώστε να αποτελέσουν την ε, ήρεμη δύναμη η οποία θα μπορέσει να συνεισφέρει. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνολική προσέγγιση και από πλευράς ΝΑΤΟ και πολλές φορές ε, ε, πρόκειται για παρεξήγηση θεωρούν ότι αυτή η συνεκτική προσέγγιση θα συνδέσει το στρατιωτικό σκέλος και πολλές φορές το ΝΑΤΟ ζητά να έχει ανοιχτό διάλογο ε, με μας. Έμπρακτα θα το δούμε αυτό. Ορισμένα γενικά σχόλια ως προς την ΕΙΕΔ και την ανθρωπιστική βοήθη. Η ΒΟΗΣ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκαν υπέρ του ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να είναι εκτός ε, ε, δράσης και εντολής της ΕΙΕΔ, διότι ε, δεν σχετίζεται με όλες τις πτυχές της ΚΕΠΑ. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για τον κώδικα συμπεριφοράς του ICRC που θεωρεί ότι οι δωρητές θα πρέπει να χορηγούν αυτονόμως ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι ένα μέσο διαχείρισης κρίσεων. Τα τρία θεσμικά όργανα υπέγραψαν αυτό το πλαίσιο του 2009. Αν κοιτάξουμε το ε, παρελθόν αλλά και το μέλλον ως προς, τα, ως προς θέατρα επιχειρήσεων θα πρέπει να δούμε κατά πώς θα υπάρξει αντίσταση σε αυτή τη συνεκτική προσέγγιση. Η ΕΕΔ δεν θα πρέπει να εντάξει την ανθρωπιστική βοήθεια στους άλλους τομείς, στη γενικότερη της δράση δηλαδή. Ως προς την ε, παρούσα κρίση της Λιβύης, το Συμβούλιο στα συμπεράσματα στις 30 ε, Μαρτίου θεώρησε ότι η ΚΕΠΑ θα πρέπει να ανταποκριθεί και στις ανθρωπιστικές ανάγκες σύμφωνα με την εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Το μόνο που θα μπορούσε, επί το οποίο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη θα ήταν ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές, το στρατιωτικό σκέλος είναι και το τελευταίο. Είναι το μέσο τελικής προσφυγής. Υπάρχει όμως κάποια σύγκυση στα μέσα και σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις και δεν υπήρξε ένα τέτοιο αίτημα ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη. Όμως τα κράτη-μέλη στα συμπεράσματα έλαβαν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία, δηλαδή το ε, αίτημα της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας και θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η σύμπραξη εάν τύχει καλής διαχείρισης και εποπτείας, καθώς και αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως να υπάρχει κοινή αποδοχή και από τα δύο μέρη. Χαίρομαι που ο κύριος Νιώτσο είναι εδώ, διότι θα μιλήσουμε και μέσα στα πλαίσια του, της μονάδας διαχείρισης καταστάσεων κρίσης. Μας μιλήσατε για το νέο σας ρόλο χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα πλατφόρμα για την ύπατη εκπρόσωπο έτσι ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί με όλες τις αρμοδιότητες, επιμέρους αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι δεν θα υπάρχει επικάλυψη με την ΕΚΟ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας, αλλά θα δούμε ποια θα είναι η εντολή σας έμπρακτα ως προσμένες συστάσεις και ρήτρες διαφύλαξης. Κατά την άποψή μας, η εντολή της ΕΚΟ ως προς το πολιτικό σκέλος είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης της ΕΚΟ με τα άλλα μέσα. Επειδή υπάρχει σύγχυση και όχι σαφής οριοθέτηση, θα πρέπει να συζητήσουμε με την Ε.Ε.Δ. και τα κράτη-μέλη για την εξισορρόπηση των μέσων, για την ανταπόκριση, την ανθρωπιστική ανταπόκριση. Ξέρουμε ότι... Γνωρίζουμε ότι η δική σας πλατφόρμα δεν είναι αποκλειστική και θα θέλαμε να μας πείτε ποιους θα πρέπει να συμβουλευτούμε στην ΕΙΕΔ ως προς ε, τις κατευθυντήριες γραμμές είναι απόλυτα σαφής για το ανθρωπιστικό, ως προς το ανθρωπιστικό χάσμα που θα πρέπει να καλύψουν οι στρατιωτικές δυνάμεις όταν δεν υπάρχει πολιτική εναλλακτική λύση για να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για την χορήγηση της βοήθειας θα πρέπει να υπάρχουν μέσα συντονισμού μεταξύ ΕΙΕΔ και ΕΚΟ από όλα τα επίπεδα, από την ύπατη εκπρόσωπο μέχρι την ε, Κομισιόν στο σύνολό της. Θα πρέπει να μην υπάρχουν επικαλύψεις με την εντολή της ΕΚΟ. Αυτό ε, καταγράφεται και στις συνθήκες. Τώρα, ως προς μία κατανόηση της όλης δράσης στην ΕΙΕΔ ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια που αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας μας, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τηρήσουμε αυτές τις αρχές. Ορισμένα συμπερασματικά σχόλια. Δυστυχώς υπάρχει σύγχυση ρόλων και αυτό φάνηκε και στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει να ζήσουμε αυτό. Πώς μπορούμε όμως να ελαχιστοποιήσουμε την επιπρόσθετη ενδεχόμενη ζημία. Αυτό είναι το ουσιώδες. Η πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και την απτυξιακή βοήθεια. Γιατί και εκεί υπάρχει πολιτικοποίηση. Ίσως η Ε.Ε. αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβάλλει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην συνεκτική, δηλαδή ως προς τις ανθρωπιστικές αρχές και τους ανθρωπιστικούς παράγοντες, έτσι ώστε να έχουμε σταθεροποίηση και σωστή διαχείριση κρίσης για να καταβάλουμε προσπάθειες η οικοδόμηση της ειρήνης και να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρτίνες. Ο κύριος Ζάγκελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που οργανώνετε αυτό το πάνελ. Η ακρόαση αυτή είναι άκρος σημαντική. Πριν αρχίσω μπορώ να πω ότι δέχομαι τις περισσότερες παρεμβάσεις και εάν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν είμαι, εγώ τουλάχιστον ερωτήματα δεν είμαι καθόλου ε, ανήσυχος ως προς τις ε, κατευθυντηρίες γραμμές μας. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το τι μιλάμε. Όταν μιλάμε για πολιτικοποίηση θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει. Όταν μιλάμε για στρατιωτικοποίηση θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η διαφορά, όπως είπε και ο κύριος Mountain. Δηλαδή μιλάμε για στρατιωτική επέμβαση καθαρά υποστηρικτική για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ανθρωπιστικών φορέων. Αυτό είναι κάτι το οποίο εφήγει σήμερα το πρωί από όλους, όμως θα πρέπει να προβαίνουμε σε διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου όπως το Αφγανιστάν, όπου, όπου οι στρατιωτικοί ανέλαβαν και τον, ε, το ανθρωπιστικό αυτό έργο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή το περιεχόμενο ανθρωπιστικό και η βοήθεια είναι ανθρωπιστική. Είναι σαφές και είναι απαραίτητο να τηρούμε τις ανθρωπιστικές αρχές. Διαφορετικά δεν πρόκειται για υποστήριξη και γι' αυτό μιλάμε και για ουδετερότητα των στρατιωτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν την ανθρωπιστική αυτή ε, επέμβαση, ας το πούμε. Μία υποστήριξη η οποία αφορά και το στρατιωτικό σκέλος πολλές φορές όχι τόσο στο θέατρο επιχειρήσεων, αλλά στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ έγκυται η υποστήριξη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τη διαφορά μεταξύ διαχείρισης και απάντησης σε καταστάσεις κρίσης. Εγώ δεν ασχολούμαι με, ε, με τα πολιτικά διέξοδα μίας κρίσης, αλλά την αποφυγή κρίσεων. Ως προς το γενικότερο υπόβαθρο αυτών για τα οποία θα μιλήσω, γνωρίζουμε πως έχει κατάσταση και όσο πιο περίπλοκη είναι, τόσο θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος κάνει τι. Και θα πρέπει να το γνωρίζουμε εξάντε. Δηλαδή να γνωρίζουμε ποιος θα κάνει τι αύριο, σε ποιο είδος κρίσης και στη συνέχεια Εάν η ανθρωπιστική βοήθεια θεωρηθεί πολιτικοποιημένη, θεωρηθεί και το τονίζω αυτό, είτε από τους αποδέκτες είτε από τα συμβαλώμενα μέρη, θα πρέπει να τους πείσουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διαφορετικά περιπλέκουμε τα πράγματα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο είναι ουδέτερες και αμερόληπτες αυτές οι δυνάμεις, έτσι ώστε να είναι αποδοτική και η βοήθεια. Εάν μας θεωρούν πολιτικοποιημένους, δεν μπορούμε να δράσουμε ανθρωπιστικά. Παρεμποδίζεται το έργο μας. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ναι, υπάρχει κίνδυνος. Από πού προέρχεται ακούμε ότι προέρχεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, από τη νέα ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί η νομική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ε, συνάδει πλήρως με το ανθρωπιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, όπου συμμετέχουμε όλοι όλα τα κράτη-μέλη, άρα θα ήταν αδιανόητο να ισχύει κάτι τέτοιο. Και όπως ορίζεται και από τη συνθήκη γνωρίζουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για τη συνθήκη δεν έχουμε δίκιο γιατί υπάρχουν δύο συνθήκες. Η συνθήκη για την Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της, Ένωσης. της Ένωσης. Ως προς συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα νέο άρθρο το οποίο δεν προϋπήρχε είναι το 214 που ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια και που ορίζει τις θεσμικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπενθυμίζει τις αρχές. Αυτά τα δύο στοιχεία ε, σημαίνουν το εξής ότι είναι αδιανόητο να είναι πολιτικοποιημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο στη νομική της βάση. Αυτό θα ήταν λανθασμένο εξορισμού. Η συνένεση τηρείται από όλους και προτρέχει ως προς το άρθρο 214, διότι το άρθρο 214 υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και ισχύει από τη διαδικασία κύρωσης και μετά. Μιλάμε λοιπόν για την τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων ε, Εθνών και το MCDR. Από πού προέρχεται ο κίνδυνος. Αν δεν προέρχεται από το θεσμικό επίπεδο, προέρχεται από την, ε, σχετίζεται με την επιτυχία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτοί που την αμελούσαν στην αρχή βλέπουν ότι είναι αρκετά δελαστική και αν δείτε την ατζέντα μας βλέπετε ότι ότι υπάρχει έμπρακτα βοήθεια ως προς αυτούς που αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση. Ήδη διασαφήνισα ε, το, γεγονός ότι με βάση τις αρχές μας προβαίνουμε και στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι ορίζουμε τις ανάγκες και σημαίνει επίσης ότι ο πολιτικός κόσμος αποφασίζει, μάλλον η, η κοινωνία των πολιτών αποφασίζει πού θα διανεμηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και όχι πολιτικές αρχές, τουλάχιστον δεν θα έπρεπε. Άρα, δεν έχουμε μια κατάσταση τύπου Αφγανιστάν. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε, γιατί τότε δεν πρόκειται για αμυγή ανθρωπιστική βοήθεια και το Αφγανιστάν θα θεωρηθεί μία περίπτωση αποτυχίας ε, ως προς την ανθρωπιστική, διότι δεν ήταν καθαρά ε, ανθρωπιστική, αμυγός ανθρωπιστική αυτή η βοήθεια. Άρα θα πρέπει να εξηγήσουμε στον εξωτερικό κόσμο ότι δεν είμαστε ε, δογματικοί γιατί θέλουμε να τηρήσουμε ορισμένες αρχές. Οι αρχές έχουν λόγο ύπαρξης έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτικοποίηση. Και έτσι θα πρέπει να παράσουμε τη βοήθεια. Το Αφγανιστάν μας έδειξε μία διαφορετική πραγματικότητα. Αυτό είναι το παράδειγμα που μας ε, ορίζει το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Στην πρόσφατη κρίση θα πρέπει να δούμε τι θα ε, γίνει με το Πακιστάν και με την Λιβύη. Για το Πακιστάν Νομίζω ότι βοηθήσαμε και ως προς το στρατιωτικό σκέλος μέσα στα πλαίσια της έκτακτης έκρεθμης κατάστασης ως προς τις πλημμύρες. Στο βορρά έχουμε εκτοπισμένους και πρόσφυγες και προσπαθήσαμε να κάνουμε καλή χρήση και του στρατιωτικού σκέλους. Τώρα, ως προς τη Λιβύη, αφήνω την απόφαση που ελήφθη ως προς το στρατιωτικό σκέλος. Θα δούμε πώς θα επικεντρωθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θα δούμε τι θα γίνει με τον επαναπατρισμό αυτών των ανθρώπων και την προστασία τους. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο επαναπατρισμός να γίνει βεβαίως και με την ε, στρατιωτική συνιστόσα και με το στρατιωτικό σκέλος και με τη συμμετοχή του δηλαδή. Θα μιλήσουμε και για την κατάσταση στο Τσάντ. Θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί θα πρέπει να ε, μην είμαστε δογματικοί. Εάν δεν τηρήσουμε συγκεκριμένες αρχές, σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχει πια ανθρωπιστική βοήθεια. Ή ίσως θα υπάρχουν άνθρωποι που ο καθένας με το δικό του τρόπο θα συνεισφέρει και θα βοηθά, αλλά δεν θα πρόκειται για αμυγή ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συνεχής διάλογος, όχι μόνο με την ΕΙΕΔ, στα πλαίσια μιας συνέχειας για το τι πρέπει να κάνουμε, Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι στην επιχείρηση Λιβύη, αν μπορώ να ε, μιλήσω κάπως σχηματικά, η βοήθεια αυτή, η ανθρωπιστική, ήταν εξαιρετική, που δείχνει ότι οι δύο αυτοί διαφορετικοί κόσμοι έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν. Και από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα και να θέσουμε έναν κοινό παρονομαστή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ζάγκελ. Ο κύριος Μιώτσου έχει το λόγο. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. ετοίμασα μια παρουσίαση για την ακρόαση αλλά όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές θα μιλήσω και εγώ για τα διδάγματα. Επιστρέφω από ένα ταξίδι στη Λιβύη όπου πήγα τρεις φορές το περασμένο μήνα και θέλω να μιλήσω για κάποια διδάγματα από την επιχείρηση και την κρίση στη Λιβύη. Μέχρι τώρα τι μάθαμε. Μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω. Η κρίση της Λιβύης παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης όπου υπάρχει ο κίνδυνος υπερκα... επικάλυψης ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας, την πολιτικοποίηση της βοήθειας. Μια χαρακτηριστική κρίση όπου παρουσιάζεται η σύγχυση αυτή των ρόλων είναι μια κρίση που δεν έχει επιληθεί και που μπορεί το σκηνικό να αλλάξει μέσα σε ώρες από την επίλυση της κρίσης σε στασιμότητα και στο χειρότερο σενάριο όπου η στρατιωτική επέμβαση μπορεί να καταστεί απαραίτητη για να υποστηριχθεί να υποστηριχθούν ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως είπε και ο Πίτερ Τσάγκλ, μέχρι τώρα έχουμε εξισορροπήσει τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον ε, οι Ευρωπαίοι το έχουν κάνει αυτό στη Λιβύη. Πριν από ένα μήνα όταν άρχισε η κρίση, το βασικό πρόβλημα ήταν να υποστηρίξουμε την κένωση των Ευρωπαίων και των υπηκών τρίτων χωρών από τη Λιβύη προς την Ισία και Αίγυπτο. Η ΕΚΟ ανέλαβε δράση. Επίσης ε, στρατιωτικά υποστηρίχθηκε η επιχείρηση και διευκολύναμε όλη αυτή τη δράση παρέχοντας όλη την υποστήριξη, παρέχοντας μέσα διευκολύνσεις που μπορούσαμε. Η κρίση συνεχίστηκε και τώρα επικεντρωνόμεθα μετά την ε, κένωση πάνω από 400 πάνω από ε, άνω των 400.000 που πήγαν ε, στην Τινησία και την Αίγυπτο και μετά σε τρίτες χώρες ε, χάρη στον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και τον Ερυθρό Σταυρό κλπ. Τώρα επικεντρωνόμεθα στην εσωτερική κρίση. Όπως ξέρετε η Λιβύη είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, το δυτικό που ελέγχεται από τον Καντάφη και την Κυριναϊκή ε, που ελέγχεται από το Μεταβατικό Προσωρινό Συμβούλιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Υπάρχουν εστίες κρίσης εκεί όπου είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες όπως στη Μισράτα και όταν πήγα στη Βενγάζη πριν από μία εβδομάδα υπήρχε η αίσθηση ότι κάτι δραματικό συνέβαινε στη Μισράτα. Ήταν έντονη η αίσθηση. Ευτυχώς είχαμε και από τον Ερυθρό Σταυρό και ε, στοιχεία ότι η ανθρωπιστική βοήθεια μπόρεσε να φτάσει στην πόλη. Μας είπαν ότι υπάρχει κρίση, υπάρχουν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, αλλά καταφέρνουν να δώσουν φαρμακευτικό εξοπλισμό, να πάνε οι γιατροί εκεί, να παρασχεθεί κάποια υποστήριξη. Προφανώς πρόκειται για κρίση, υπάρχουν, ε, γίνονται μάχες, υπάρχουν οι ελεύθεροι σκοπευτές, αλλά η κατάσταση μοιάζει με μια κρίση η οποία δεν επιβάλλει τη, τη χερσαία επίθεση και επέμβαση. Ξέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει αυτού του είδους την υποστήριξη. Η κυρία Άστον είπα ότι εκπρόσωπος είναι σε στενές συνομιλίες με το Διεθνή Συντονισμό από τον ΟΗΕ της Βοήθειας και είναι έτοιμο το σύστημα να παράσχει και στρατιωτική υποστήριξη πέρα από την ανθρωπιστική αν ε, χειροτερέψει η κατάσταση. Μέχρι τώρα θεωρείται ότι καλύπτονται οι ανάγκες μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια, χωρίς στρατιωτική, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε τη στρατιωτική επέμβαση. Είναι πολύ ευμετάβλητη η κατάσταση. Ο στρατός του Καντάφη άλλαξε τακτική. Τώρα στην Ασραμπίγια που είναι κοντά στην πρωτεύουσα, μια μικρή πόλη, κοντά στη Βεντάζη. Είναι σε απόσταση 200 χιλιόμετρων. Μπορούν σε λίγες ώρες να φτάσουν τα στρατεύματα του Γκαντάφη στη Βενγάζη. Δεν κινούνται με τάγκς, αλλά με τετράτροχα, τε, ε, τετρακινητήρια οχήματα ελαφρά. Είναι καινούργιες αυτές οι στρατιωτικές τακτικές και μπορούν να αλλάξουν ε, δραματικά την κατάσταση ακόμα και στην Βενγάζη. Ε, όπου ισχύει από τον ΝΑΤΟ για απαγόρευση των πτήσεων. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι εν πάση περιπτώσει. Και ζητήσαμε να είναι έτοιμες οι δυνάμεις να επέμβουν. Η επέμβαση θα γίνει βέβαια οπωσδήποτε με βάση το αίτημα από την Ηνωμένα Έθνη και την ΟΤΣΑ. Μέχρι τώρα ε, επικουρούμε σε μια κατάσταση όπου δεν παρατηρείται μείζον ανθρωπιστική κρίση, τουλάχιστον στην Ανατολική Λιβύη. Το δυτικό τμήμα της χώρας εξακολουθεί να ελέγχεται αρκετά στεναρά από τον Καντάφη και η ανθρωπιστική βοήθεια προσπαθεί να φτάσει το σκοπό της, ακόμα και η αποστολή του ΟΗΕ επιχειρεί να φτάσει στην Τρίπολη και να ξαναρχίσει να εργάζεται από την Τρίπολη, με βάση την Τρίπολη για να καλύπτει το δυτικό τμήμα. Στηρίζουμε τις προσπάθειες, είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΚΟ θα συνεχίσει να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να στηρίξουν το Ηνωμένα Έθνη και τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Για να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση, νομίζω ότι η κρίση στη Λιβύη είναι καλό παράδειγμα καλής διαχείρισης. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν συνεχίσουμε να επιχειρούμε όπως μέχρι τώρα, η κρίση στη Λιβύη θα αποδείξει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα συνεχιστεί, θα μπορεί να συνεχίζεται σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές. Θα πρέπει σε πολιτικό επίπεδο να στηρίξουμε την ανοικοδόμηση, ο προσωρινό συμβούλιο, να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και τον κόσμο που θα θέλει ε, απελπισμένα να αλλάξει μετά από 42 χρόνια εξουσίας του Γκαντάφη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα περάσουμε στις ερωταποκρίσεις. Έχουμε χρόνο. Υπάρχει κατάλογος. Θα δώσουμε το λόγο σε όσους τον ζήτησαν. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές που καταπιάστηκαν με πολύ σημαντικά θέματα ε, νομίζω ότι το κλειδί είναι το Αφγανιστάν όμως θεωρώ. Υπάρχει μια σημειολογική διαφοροποίηση, δεν ξέρω αν την έχετε αναλύσει. Η πολιτική, η στρατιωτική είναι καινοτόμη και δημιουργική προκειμένου περί της στρατιωτικής ορολογίας. Αντί για πόλεμο λέμε αποστολή σταθεροποίησης ή πριν από δύο εβδομάδες δεν μιλούσε κανείς για βομβαρδισμούς αλλά για εξουδετέρωση του βαρέως οπλισμού που θα μπορούσε να απειλήσει τους άμαχους. Εξουδετέρωση, ουδετεροποίηση βαρέως οπλισμού που θα μπορούσε να απειλήσει τους αμάχους. Αυτό ακούγεται καλύτερα από βομβαρδισμούς, από, από τη βομβαρδισμή. Έχουμε πληθώρα καινούρια ορολογία. Ξαφνικά οι στρατιωτικοί άρχισαν να διοργανώνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για τους πολίτες, για τους άμαχους και μιλούν για ανθρωπιστική βοήθεια η οποία παρέχεται μέσα από στρατιωτικούς φορείς. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Βεβαίω το περιεχόμενο είναι η βοήθεια. Τι βοήθεια όμω είναι αυτή, δεν είναι ανθρωπιστική με την κυριολεκτική έννοια τη λέξη. Δεν ξέρω λοιπόν αν πρόκειται μάλλον για στρατιωτική βοήθεια. Αν μιλήσουμε για βοήθεια, ίσως θα πρέπει να βρούμε μια ορολογία, μια έννοια, η οποία θα οριοθετεί το έργο των στρατιωτικών σε αντιπαράθεση με την ανθρωπιστική βοήθεια, ώστε να μην γίνει πολιτικοποίηση, να μην ε, υπησέλθει ο στρατιωτικός φορέας την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά πρέπει να οριοθετήσουμε τι είναι πολιτική επιχείρηση, τι είναι ε, στρατιωτική και τι ανθρωπιστική. Ευχαριστώ. Merci, Madame la euh, I think I couldn't agree more when uh, Peter Zangel says that Afghanistan... Ευχαριστώ. Το Αφγανιστάν είναι πραγματικά υπόδειγμα της αποτυχίας, δηλαδή της ανάγκης, της απόλυτης ανάγκης να παραμείνει ανεξάρτητη και μη πολιτικοποιημένη η ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ ήμουν στο μόνο ψυχιατρικό άσυλο του Αφγανιστάν Πήγα και το επισκέφθηκα μαζί με μια ομάδα από την Κομισιόν και ξαφνικά εμφανίστηκαν ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, πολύ καλοί άνθρωποι, που ήθελαν να αναδομήσουν το ψυχιατρίο και αυτό είναι παράδειγμα σύγχυσης των δύο επιπέδων. Γιατί τη στιγμή που αυτοί έχτιζαν και ξανάχτιζαν το ξενοδοχείο έγινε προσπάθεια αυτοκτονίας κάποιου τροφίμου του. Το ερώτημά μου όμως δεν αφορά αυτά. Τις περασμένες εβδομάδες από τότε ας πούμε που άρχισε η κρίση στη Λιβύη έχουμε περίεργες πληροφορίες ως προς το ποιος είναι ο υπεύθυνος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι η εξωτερική υπηρεσία. Ποιος στην Ευρώπη είναι ο Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια ο υπεύθυνο. Αν δεν θέλουμε να συγχυστούν τα επίπεδα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η κυρία Γεώργιεβα είναι υπεύθυνη και κανείς άλλος. Θα ήθελα να αποσαφηνιστεί αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νόζερ και μετά θα απαντηθούν τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Νομίζω ότι τα θέματα που θίξατε δημιουργούν περισσότερα ερωτηματικά από ότι δίνουν απαντήσεις, σε μένα τουλάχιστον. Αποσαφηνίσατε τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, αμεροληψία, ουδετερότητα, προσανατολισμός προς τις ανάγκες του πληθυσμού. Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να το δούμε καλύτερα. Όταν ζητεί ο λαός, ο πληθυσμός, τη στρατιωτική βοήθεια, αυτό είναι ένα σημαντικός δείκτης, μια ένδειξη σοβαρή, όπως στην περίπτωση της Βενγκάζης. Στις φυσικές καταστροφές, τσουνάμι, τα IT, ε, η συνεργασία είναι πιθανό μείγμα ή επικάλυψη ανθρωπιστικής βοήθειας, στρατιωτικής βοήθειας. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί ο στρατός ε, έχει υποδομή που μπορεί να αξιοποιηθεί όπως και στην περίπτωση της εκένωσης των προσφύγων ε, από τη Λιβύη. Αλλά τα άλλα παραδείγματα, η Λιβύη, ακτή ελεφαντοστούν, ε, Ιράκ, ε, είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι ε, εδώ υπερισχύει πάντα η στρατιωτική ε, πέμβαση. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Κάσμαρακ, θα πρέπει να προσέξουμε τη γλώσσα. Η σημειολογία των στρατιωτικών αλλάζει. Μιλάμε για soft power, ήρεμη δυναμία στρατηγική του ΝΑΤΟ. Αυτό μου δημιουργεί ένα δυσάρεστο συνέστημα, ε, ανατριχιάζω λιγάκι. Και ε, αν σκεφτώ την κυβέρνηση της χώρας μου, εκεί ε, ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός ε, υποχωρεί υπέρ άλλων όμως ε, παρουσιάστηκε στα μέσα ε, συνηγορώντας υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι επικίνδυνη αυτή η σύγχυση των ρόλων ε, ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων. Ε, παρακολούθησα την έκθεση για το Αφγανιστάν, ήρθα σε επαφή με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις για τους σκοπούς της έκθεσης και αποκόμισα ένα δίδαγμα, αν θέλετε. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις λένε πρέπει μας να ακούτε. Εμείς είμαστε οι πρώτες που φτάσαμε στη χώρα πριν από την έλευση του στρατού και θα είμαστε και εκείνοι που θα παραμείνουμε μετά την απομάκρυνση των ε, ενόπλων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν η πρόθεση είναι να δοθεί έμφαση μεγαλύτερη στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, στα πλαίσια της ε, βοήθειας. Επίσης η συζήτηση εδώ οδηγεί σε μια ομόφωνη ε, θέση ότι θα μπορούσαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας να κάνουμε καλύτερα τη συζήτηση αυτή γιατί εκεί μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο ε, για μια ανεξαρτητοποιημένη ανθρωπιστική ε, βοήθεια. Τι θέλετε να κάνουμε ως προς απαντήσεις, ε, θέλετε να μοιραστείτε το χρόνο, πώς θα ορίσουμε το χρόνο των απαντήσεων. Ποιος θέλει να αρχίσει παρακαλώ. σχετικά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τη σχέση μεταξύ της τελευταίας και της ανθρωπιστικής υπηρεσίας είναι σαφές ότι η Κρυσταλίνα Γεωργίευα είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει επικάλυψη, δεν υπάρχει διπλή δουλειά, δεν δημιουργείται κανένα τεχνικό ή πολιτικό πρόβλημα. Και η αποστολή μας, η, η επιχείρηση στη Λιβύη είναι σαφής. Πήγα τρεις φορές, ξέρω τι κάνουν οι συνάδελφοι από την ΕΚΟ, ε, είδα την συμβολή τους και την ωφέλεια που προέκυψε από αυτήν. Είμαστε στην τελευταία αποστολή όπου συζητήσαμε επί ώρες με τους συναδέλφους από την ΕΚΟ και μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα, της πληροφορίας την εικόνα από, μέσα από την ανθρωπιστική σκοπιά. Οφεληθήκαμε από τα στοιχεία αυτά και με βάση αυτά τα στοιχεία προχωρούμε εμείς στην άλλη πρωτοβουλία παράλληλα με την ανθρωπιστική πρωτοβουλία και βοήθεια για την αξιοποίηση ε, της βοήθειας που είναι μέσω σταθερότητας κλπ. Έτσι λοιπόν για μας, παρόλο που στην αρχή είχαμε κάποια προβλήματα κατανόησης του ρόλου της δικής μου της υπηρεσίας και το ρόλο της ΕΚΟ και της ανθρωπιστικής βοήθειας, νομίζω ότι τώρα όλο και περισσότερο πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να προσθέσει κανείς κάτι ίσως. Ε, oui, merci. Deux, trois points. Ε. Δύο, τρία σημεία. Όπως σας είπα, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας, λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας λειτουργεί εδώ και 15 μήνες και από την 1η Δεκεμβρίου του 2009 τηρούμε κατά γράμμα τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ως προς την ερώτηση του κυρίου Βέρμαν, η, όπως σας είπα και όπως γνωρίζετε, η κυρία Γεωργίευα ε, είναι επικεφαλής ως προς την Λιβύη. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε από την ε, αρχή και οι ενδιαφερόμενοι είναι στη Βενγάζη για να διαχειριστούν την κατάσταση, την κατάσταση αυτή. Εκεί δεν αντιμετωπίσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ε, χρειάζεται εποπτεία, αλλά ήπια εποπτεία ε, λειτουργεί πολύ καλά και είναι πολύ καλό το ότι έχουμε τους εμπειρογνώμονες εκεί για να δούμε ε, πώς έχει η κατάσταση στην ε, Τρίπολη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανθρωπιστικές ανάγκες και βεβαίως αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μαύρες ζώνες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εάν κάποτε ε, αλλάξει αυτή η κατάσταση, τότε οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΟ θα μεταβούν όπως ισχύει κατά αναλογία και στο, ε, στην ακτή του Ελεφαντοστού, όπου η κατάσταση έχει αλλάξει τις τελευταίες 36 ε, ώρες. Θα πρέπει να δούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις Λιβύη και Ακτή είχαμε προβλέψει 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί. Στη Λιβύη για τον επαναπατρισμό και στη Λιβερία επίσης για να υποδεχτούμε αυτούς που έχουν διαφύγει από την ακτή του ελεφαντοστού. Και τώρα θα γίνει το αντίστροφο για τον επαναπατρισμό. Εάν, υπάρχουν, ε, εάν υπήρχαν λόγια ανησυχίας, τώρα πια δεν ισχύουν. Νομίζω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε διότι συμβαδίζουμε με τη συνθήκη και ως προς την ε, ανθρωπιστική βοήθεια μπορούμε να πούμε ότι ανταποκρινόμαστε στην κατάσταση και χορηγούμε σωστά ανθρωπιστική βοήθεια. Και κάτι το τελευταίο ως προς τη, το στρατιωτικό σκέλος. Ο κύριος Κασμάρεκ μίλησε για σημασιολογική δημιουργία. Αυτό δεν αποτελεί προνόμιο των στρατιωτικών. Αν κάνετε μία έρευνα στο Google θα δείτε ε, υπό το λίμα ανθρωπιστική βοήθεια ότι υπάρχουν ε, οι περισσότερα, περισσότερα δεδομένα. Όταν κάποιος μου λέει ότι κάποιος χρησιμοποίησε τον ε, όρο ανθρωπιστική, ανθρωπιστικός, πάντα ρωτώ να μάθω τι εννοεί. Γιατί ο καθένας μπορεί να εννοεί κάτι το εντελώς διαφορετικό. Η κυρία Τζίμερ, 30 δευτερόλεπτα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι παρά τις απαντήσεις σας που είναι άκρος ε, καθυσυχαστικές, θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομική ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι έγιναν απόπειρε στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει πιο, να υπάρξει μια σύγχυση γύρω από την διαχωριστική γραμμή Τη ανθρωπιστική βοήθεια που αρχίζει και που σταματάει. Και στην ε, περίπτωση της Βορείου Αφρικής υπάρχουν ε, ε, πολλές φωνές που ακούγονται. Δεν αφορά μόνο την κυρία Γεωργίευα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σαφή οριοθέτηση. Θα ήθελα την γνώμη του κύριου Τζάγκλ και των δύο άλλων ε, πάνελιστ. Η κυρία Τζίμερ. Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Δεν έχω την εντύπωση ότι από αυτά που ακούσαμε οριοθετούνται οι δύο φορείς. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί ο διαχωρισμός που θέλουμε να μην μπορεί να γίνει στην πράξη και ότι προφανώς πάντα θα υπάρχουν και κίνδυνοι και επικαλύψεις και κίνδυνοι για αυτούς που συμμετέχουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Όμως ε, συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί να είναι εκεί. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δούμε εναλλακτικέ λύσεις. Δηλαδή επιχειρήσεις ε, υπό, τον, ε, υπό τα Ηνωμένα Έθνη ε, και προστασία από καταστροφές. Δυνατότητες προστασίας από καταστροφές. Όχι υπό την ευθύνη των στρατιωτικών φορέων, αλλά υπό των πολιτικών. Τι θα μπορούσε να γίνει ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ε, έχετε το λόγο, κύριε Μάουντεν. Και η κυρία Μαρτίνες θα απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω το θέμα της ε, σαφήνειας των χωριστών ρόλων. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση των διαφορετικών ρόλων ακριβώς. Το είπαν και άλλοι. Καμιά φορά βέβαια είναι δύσκολο να έχουμε σαφείς όρους, Παραδείγματο χάρη προστασία των όπλων, των αμάχων. Είναι κάτι που ενδιαφέρει όλο και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα και αν δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή για πολλά χρόνια το κύριο πρόβλημα ήταν η συνεχώς μετατοπιζόμενοι πληθυσμοί. Από τότε υπήρξε μια εξέλιξη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τώρα νομίζω ότι πολλοί, αν όχι πολλές αν όχι περισσότερες ανθρωπιστικές αποστολές του ΟΗΕ όπως στο Κονγκό έχουν ως πρώτη τους προτεραιότητα την προστασία των αμάχων. Και αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που χορηγούνται για αυτόν τον σκοπό πρέπει να τον εξυπηρετούν και αυτές. Αλλά οι στρατιωτικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι για τέτοιου είδους δουλειές και γι' αυτό Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πρόσθετη εκπαίδευση των στρατιωτικών. Δεν απαιτείται πάντοτε μόνο καθαρά στρατιωτική δράση όπως η no-fly zone, αλλά καμιά φορά ζητιέται η εφαρμογή ανθρωπιστικών προγραμμάτων όπως την παρεμπόδιση επιθέσεων. Δεν μοιράζουν οι στρατιωτικοί μεν τρόφιμα και φάρμακα, αλλά διασφαλίζουν τη χορήγησή τους από άλλους. Δεν είναι με καθαρά ανθρωπιστική δραστηριότητα, αλλά έχει ανθρωπιστικές επιπτώσεις, δηλαδή επιτρέπει στους ανθρωπιστικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Μπορεί να μην είναι σαφή όλα αυτά στην έκφρασή τους, αλλά πρέπει να τα καταλάβουμε σαφώς ποιο ρόλο παίζει ο καθένας. Οι στρατιωτικοί ως ειρηνευτές ή όχι έχουν όρια στη δράση τους. υπάρχει και άλλη σύγχυση. Μίλησαν πολύ για το Αφγανιστάν. Δυστυχώς εκεί η σύγχυση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και στρατιωτικής δράσης οδήγησε στην πεποίθηση μερικών Ταλιμπάν ότι η ανθρωπιστική είναι απλώς μία προέκταση των στρατιωτικών και αποτέλεσμα υπήρξε βέβαια πολύ αρνητικό επιθέσεις κατά των ανθρωπιστικών και φυσικά κατά των ανθρώπων που προσπαθούν αυτοί να βοηθήσουν και που γίνονται στόχοι επιθέσεων. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε γιατί οι διεθνείς δυνάμεις αυτή τη στιγμή φεύγουν από το Αφγανιστάν αλλά οι ανθρωπιστικοί πρέπει να παραμείνουν και να δράσουν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ό,τι μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη Λιβύη πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να δω ακριβώς πώς θα γίνει και εκεί η διάκριση των δύο λειτουργιών. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό όπως λέμε και εδώ, να διαχωρίσουμε τα πολιτικά συμφέροντα από άλλα. Φυσικά υπάρχει το ΕΚΟ και η ευρωπαϊκή προσέγγιση, υπάρχουν όμως και χωριστά με μονομένες χώρες μέλη με δικό τους πρόγραμμα. Και πρέπει να διαχωρίσουμε το πολιτικό συμφέρον από τα άλλα Πολλές χώρες είπαν ότι το πολιτικό του συμφέρον είναι να εγκαταλείψει την εξουσία ο κύριος Καντάφη. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα σχέση με το κατά πόσον θα βοηθηθεί η ανθρωπιστική δράση γιατί αυτή αφορά και τις ζώνες που ελέγχει ο Καντάφη. Έτσι βλέπετε πόσο μπερδεύονται τα πράγματα. Κυρία Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, για να απαντήσω, ίσως πάλι θα δημιουργήσω περισσότερες ερωτήσεις για την ορολογία, σημειολογία. Συμφωνώ για να το πω απλουστευτικά, όταν μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική, είναι σαφή η συνθήκη σε σχέση με τους στόχους της αναπτυξιακής, δηλαδή είναι η εξάλληψη της φτώχειας και μπορούμε να σημειολογικά να συζητήσουμε την φτώχεια κλπ. Αυτό που μάθαμε από το Αφγανιστάν όμως είναι ότι η εκπαίδευση, για παράδειγμα, είναι κάτι παραπάνω από το χτίσιμο ενός σχολείου δεν έχει να κάνει μόνο με τα τούβλα, αλλά την ποιότητα της εκπαίδευσης, ε, η πρόσβαση στα σχολεία, στην εκπαίδευση από τον κόσμο κλπ. Είναι συνεχιζόμενη συζήτηση, αλλά συμφωνώ βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ρόλων, επειδή είναι σαφείς και οι αρχές. Συμφωνώ, Ρώσ, με αυτό που λες σχετικά με την αντίληψη. Είναι σημαντικό αυτό στην περίπτωση του, της δικής μου οργάνωσης και άλλων. Ε, είχαμε προϋπάρξει Τη στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Είμαστε εκεί στη χειρότερη κρίση και προτιθέμεθα να μείνουμε για να συμβάλλουμε στη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση. Θέλουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη του κόσμου εκεί. Η αντίληψη λοιπόν του ρόλου μας είναι πολύ σημαντική για την πρόσβαση που θα έχουμε. Για το ρόλο των στρατιωτικών. Δεν θα μιλήσω για του εθνικού στρατου, γιατί παίζουν ρόλο στην αντίδραση σε μια κρίση όπω το Πακιστάν για παράδειγμα είναι σαφές ότι αναγνωρίζομαι ότι μπορεί οι στρατιωτικοί να παίξουν ένα ρόλο ως σύστατη λύση. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Ο τύπος της ε, βοήθειας, συνεργασία και διάλογος. Χρειάζονται 10 χρόνια για να καταλάβουν μερικοί τις συνέπειες αυτών των δράσεων. Οι συνάδελφοι που ε, ετοιμαζόντουσαν για την ακρόαση μου είπαν ότι ε, τώρα περνάνε τα μηνύματα στο Αφγανιστάν μετά από 10 χρόνια. Συμφωνώ με το διάλογο. Σε κυβερνητικέ οργανώσει θα πρέπει να αποφασίσουμε και να ε, σκεφτούμε τι είδου διάλογο θέλουμε. Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού. Πρέπει να καταλάβουμε ίσω ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμό μαζί με τους στρατιωτικούς ε, όχι συντονισμός των δικών μας επεμβάσεων. Επίσης για την ανεξαρτησία της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ακόμα μέχρι τώρα είναι ανεξάρτητος δωρητής, ε, θέλει ανεξαρτησία και ουδετερότητα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, όπως είπε και ο κύριος Τσάγκλ, μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος ε, να μην συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ΚΕΠΑ. Θα πρέπει να δούμε τις ε, ήπιες αρμοδιότητες που έχουμε εμείς, την ήρεμη δύναμη, έχουμε τους πόρους, έχουμε τον προϋπολογισμό και μιλάμε για ανθρωπιστική αλλά και ανθρωπιστική, ε, ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. δεν θα συμφωνήσουμε για μια εξωτερική πολιτική αλλά άλλες πτυχές πάλι εξωτερικών πολιτικών για να το πω ομά, οι συνθήκες είναι σαφές, σαφείς σχετικά με τους στόχους. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψε. Α, με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει, με συγχωρείτε. Ναι, και έχουμε και χρόνο. Η ερώτηση του κυρίου Μπέρμαν καταρχήν, αν υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον στη διαμόρφωση των ε, μηχανισμών της νοσιακής ε, ανθρωπιστικής βοήθειας θα μπορούσε να υπάρχει σύγχυση με άλλες. Χάρη στην σαφήνεια των μηνυμάτων από το Κοινοβούλιο και από την Επίτροπο ε, που ανέφερε στο Λονδίνο την έκφραση «over my dead body» ότι εδώ πιστεύουμε ότι θα παραμείνει για καιρό η βοήθεια αυτή. Το πρόβλημα τέθηκε, αλλά απαντήθηκε. Η ερώτηση της κυρίας Τσίμερ. Πάντα μπορούμε να διαβάσουμε διάφορα κείμενα, να τα ερμηνεύουμε ανάλογα με τις προτεραιότητές μας. Σε ό,τι αφορά την απόφαση για τη Λιβύη, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι και η αιτιολογική σκέψη 5 και το άρθρο 1 σαφώς ε, αναδεικνύουν δύο στοιχεία, όπου το ένα είναι ότι πρόκειται για υποστηρικτικό μέτρο αυτό που προγραμματίζεται από τη U4 προς την, ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια και δεύτερον είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται όχι μετά από αίτημα των Ηνωμένων Εθνών αλλά της ότσα, ούτως ώστε να ε, υπάρχει αυτή η πολιτική και ανθρωπιστική διάσταση. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο και αυτό που είδαμε και από τη Βαρόνη Άστον ευθυγραμμίζεται με αυτή τη βασική αρχή. Επίσης για την πολιτική προστασία και αν εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, όπως ξέρετε τον Οκτώβριο ε, είχαμε κάνει μια σχετική ανακοίνωση που συνολικά είχε θετική απήχηση. Το Κοινοβούλιο ασχολείται ακόμη με τη γνωμοδότηση και πιστεύω ότι θα είναι υποστηρικτική. Ε, ίσως είμαστε αρκετά μετριοπαθείς ε, ακόμα στην Κομισιόν, αλλά θα πρέπει πάντοτε να ε, σταθμίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε Τώρα είμαστε στο μέσον της διαδρομής. Οπωσδήποτε στην πολιτική προστασία καλό είναι να ε, βοηθηθούμε αν είναι δυνατόν. Αλλά δεν συμφωνούν, δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος όλα τα κράτη-μέλη. Και το καλοκαίρι θα ε, καταρτήσουμε και αργότερα θα υποβάλλουμε τα σχετικά κείμενα. Επίσης, όταν συζητήσουμε για τις νομικές βάσεις, θα έχουμε πάλι μια μεγάλη ευκαιρία να επανέλθουμε στη συζήτηση όλων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα να έρθουν οι τρεις επόμενοι ομιλητές. Θα μιλήσουμε για την διαχείριση της σχέσης στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους ε, και θα μιλήσουμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Διακόπτουμε για δύο λεπτά. Monsieur Caramba, Καμπάμπα, Κανάσα,

Donc, euh, nous avons le Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε κύριο Καμπάμπα από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης που θα μας μιλήσει για την περίπτωση της λαϊκής ε, δημοκρατίας του Κόγκο και θα μας μιλήσει για την αποστολή του για τη διατήρηση της ειρήνης. Μετά τον, θα ακούσουμε τον κύριο Γκανάσα, ο οποίος ασχολήθηκε ε, με την περίπτωση του Τσάντ και της ε, Δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής και μετά την κυρία Ίγκριτ Μακδόναλτ που είναι υπεύθυνο ε, της εκστρατείας υπέρ των προσφύγων στην Νορβηγία. Θα έχετε το λόγο για 8 λεπτά ο καθένας. Κύριε Καπάμπα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. θα ήθελα να σας πω ότι μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια αφενός και για τη στρατιωτική σκέλος. Το Νοκούντα Μοτζόμπ είναι μία έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε το 2008 κατά την ε, κρίση. Κούντα Πρόκειται για έναν στρατηγό ο οποίος ξυλώθηκε από τη θέση του και, ε, και δημιούργησε ένα δικό του, μη δική του ε, μονάδα. Γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση «no kunda, no job». Δηλαδή τη στιγμή που δεν υπάρχει ο κούντα δεν υπάρχει και, και εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το στρατηγικό σχέδιο, το ιδεολογικό και το οικονομικό αυτής της ε, βάσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι ότι όταν δούμε τους διάφορους φορείς που δρούν επί οποίο, ο Κούντα δημιούργησε αυτή την, ε, την μονάδα, αυτό το Αντάρτικο και βλέπουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συνεργασία με την κυβέρνηση του Κονγκό σε περίπτωση και φυσικών καταστροφών και έκτακτης έκρηκμης αριθμιστικής ανθρωπιστικής κατάστασης για να δούμε τι ε, μπορεί να γίνει με την ε, χρήση των φυσικών πόρων όπως των μεταλλευμάτων. Στην περίπτωση του no kunda no job μπορούμε να δούμε τι εμπίπτει στο κεφάλαιο 7. Πρόκειται για την, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών μέσα στα πλαίσια του κεφαλαίου 7 και την προστασία των αμάχων. Όταν μιλάμε για προστασία των αμάχων και όταν μιλάμε για καταστροφές, μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια. σε σχέση με τον στρατό του Κονγκό, ο στρατός του Κονγκό δεν είναι καλά διαρθρωμένος και δεν μπορεί να αντισταθεί στις άτακτες δυνάμεις του ε, Κούντα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιταχθεί στους αντάρτες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία σταθεροποίηση προς Ανατολάς της χώρας. Υπάρχουν, υπάρχει και η πολιτοφυλακή Μάι που είναι ένας άλλος παράγων. Φτάσαν πολλοί πρόσφυγες από παντού, πολύ εκτοπισμένοι και έτσι η πολιτοφυλακή μπόρεσε να λαιλατήσει αυτούς, ε, αυτούς τους ανθρώπους και πρόκειται και για ένα φυτόριο για να μπορέσει να στρατολογήσει πολλά παιδιά για μελλοντικές σειράξεις. Το ζήτημα λοιπόν σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια και τους ανθρωπιστικούς διεθνείς φορείς είναι να δούμε τι συμβαίνει επί το οποίο και πώς μπορούν οι διεθνείς οργανώσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση στους εκτοπιστέντες, πρόσφυγες και πώς μπορούν να βρουν ένα διάβλο για να δώσουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια. Προς Ανατολάς βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί εκτοπιλισμένοι, μεταφέρονται πολλοί, οι οποίοι την χάνουν της προστασίας των Ηνωμένων Εθνών. Από τους κιανόκρανους δηλαδή. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτή την τάση. Ιδεολογικά συνειδητοποιούμε ότι όταν μετατοπίζεται ο πληθυσμός και όταν υπάρχει μεγάλη παρουσία προσφύγων, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο ανατολικό μέτωπο της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Δηλαδή χρειάζονται όχι μόνο ανώκρανοι, αλλά και άλλες διεθνείς δυνάμεις. Η διεθνής βοήθεια ορίζεται και ως προς το οικονομικό της σκέλος. Με την μεγάλη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούμε να ε, παράσχουμε τρόφιμα σε πολλά εμπορικά κυκλώματα και αυτό σε τοπική βάση. Αυτή η μετατόπιση πληθυσμών προς τους καταβλισμούς θα πρέπει να εξασφαλιστεί υπό τις, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, κάτι το οποίο δεν ισχύει, διότι πολλές φορές λαιλατούνται τα αγαθά αυτών των πληθυσμών και στην, ε, στο ψήφισμα 1925 των Ηνωμένων Εθνών προβλέπεται η προστασία από τους ε, κιανόκρανους. Μετά το 2008, δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την προστασία των πολιτών, των αμάχων. Το 2008 μιλάμε για 1.200.000 εκτοπισμένους, εκατοντάδες χιλιάδες ε, νεκρούς και δυστυχώς ε, δεν μπορέσαμε να ε, αντιμετωπίσουμε αυτή την έκρηκνη κατάσταση λαϊλασίας. Όταν μιλάμε για στρατιωτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, θα πρέπει να αναφερθούμε στο Κονγκό ιδιαίτερα, διότι τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να προστατεύσουν τους πολίτες και τους αμάχους, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους αντάρτες και τα διάφορα αντάρτικα για να μην μπορέσουν να πλήξουν αυτές τις περιοχές και τους αμάχους. Τι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί εν κατακλείδη. Θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά τα Ηνωμένα Έθνη όταν μιλάμε για προστασία αμάχων. Θα πρέπει να έχουμε πολεμικές σειράξεις για να προστατεύσουμε τους πληθυσμούς. Οι οικιανόκρανοι μπορούν να προστατεύσουν τους αμάχους. Εδώ δεν έχουμε σαφείς απαντήσεις από νομικής πλευράς και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο το κεφάλαιο 7 των Ηνωμένων Αθνών είναι απόλυτα σαφές. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι άμαχοι πλήττονται ιδιαίτερα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο στρατηγός Γκανάσα έχει το λόγο. Ήμουν στρατηγός, γιατί τώρα είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος. Και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που ζητούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ως προς τον διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικών και ανθρωπιστικών οργανισμών. Και τώρα ασχολούμαι με έναν οργανισμό που αφορά την οργάνωση υπηρεσιών ασφαλείας. Είναι ενδιαφέρον ότι με καλέσατε εδώ. Εμένα η παρουσίασή μου λέγεται ο ανθρωπιστικός χώρος και η ελευθερία της στρατιωτικής δράσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι μία πτυχή που παρέμεινε στη μνήμη των ανθρώπων ε, στο πρόγραμμα παρέμβασης στο Τσάντ ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια που προσπαθήσαμε να χορηγήσουμε στα Ανατολικό Τσάντ σε συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η επιχείρηση αυτή χαρακτηρίστηκε από το εξής παράδοξο που οφείλεται στον πολύπλοκο χαρακτήρα της. Η εντολή μας αφορούσε την προστασία του πληθυσμού, αλλά χωρίς την άδεια να παρεμβληθούμε μεταξύ Τσάντ και Σουδάν. Η επιχείρησή μας λοιπόν ήταν προσωρινή μέχρι να εμφανιστεί μια δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά την οποία δεν ήθελε το Τσάντ. Η Ευρώπη θέλησε να ενισχύσει την πολιτική ασφαλείας της, αλλά η κύρια χώρα που έστειλε δυνάμεις εκεί η Γαλλία ήταν δεμένη στο τσάντα από συμφωνίες που προϋπήρχαν. Υπήρχε και το πρόβλημα των ληστών που ήταν οργανωμένοι σε εθνοτική βάση. Τέλος η κυβέρνηση του Τσάντ είχε δεχτεί την ανάπτυξη αυτής της ξένης δύναμης μόνο και μόνο γιατί ανέμενε πολιτική και στρατιωτική επίπτωση αλλά όχι τη βελτίωση της ζωής του πληθυσμού του. Σε αυτό το περίεργο πλαίσιο αναπτύξαμε τις προσπάθειές μας και έτσι κάναμε τις πρώτες επαφές με, με, ανθρωπιστικές με οργανώσεις. Λέω ότι ήταν περίεργο αυτό διότι οι επαφές ήταν μεν πολύ θετικές και θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μία απλή και αποτελεσματική σχέση που και στους θεωρητικούς τους όρους ήταν απλή προστασία, προστασία, προστασία των πληθυσμών που θεωρούνταν ευάλωτοι όπως οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί, περίπου 400.000 άνθρωποι με 4.000 στρατιώτες συνοδεία σε ένα έδαφος σαν τη μισή Γαλλία. Προστασία των ανθρωπιστικών, 2.000 άνθρωποι που εκπροσωπούσαν καμιά δεκαριά οργανώσεις με διαφορετικές πολιτικές θέσεις και καθεστώτα και τέλος προστασία των τοπικών πληθυσμών που εκτίθενταν σε επιθέσεις. Στα λόγια απλά όλα αυτά, αλλά στην πράξη πολύπλοκα. Θα μπορούσαν να ήταν απλές οι σχέσεις εφόσον είχε υποθεί ρητά ότι η αποστολή μας που ήταν κυρίως στρατιωτική αν και αδέκαστη δεν λέω ουδέτερη εφόσον όλα αυτά είχαν αποδειχθεί δηλαδή χωρίς συνεργασία του πολιτικού με το στρατιωτικό σκέλος δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα για να κατακτήσουμε τις καρδιές των πληθυσμών και οι επιθέσεις των εξεγερμένων χειροτέρευαν την κατάσταση αισθητά. Τα λογιστικά προβλήματα ήταν σχεδόν ανυπέρβλητα. Τότε ο κύριος Κουστέρ πήγε στο Τσάντ το Φεβρουάριο και είχε πει μπροστά στους ανθρωπιστικούς ότι πρέπει να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να προστατευτούν οι εκτοπισμένοι πριν από την εποχή των βυροχών η δήλωση εκείνη δημιούργησε ένα δίλημα για μας τους στρατιωτικούς. Διότι απ' τη μία αν δεν θεωρούσα τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ως καθαρά εφαρμόσιμες άμεσα, απ' την άλλη δεν μπορούσα και να τις αγνοήσω λόγω των πολιτικών σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ Τσάδ και Γαλλίας ή Ευρωπαϊκής Ένωσης που τότε προεδρευόταν από τη Γαλλία. Η υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ είχε υπολογίσει ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των εκτοπισμένων, των, εκτο, των μετατοπιζομένων, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει οτιδήποτε απτό για να αυξηθεί η ασφάλειά τους. Τέλος, λόγω της βίαιης ρήξης των σχέσεων με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, Oxfam και άλλες, χρειάστηκε να πάρω κάποια απόφαση. Θεώρησα σωστότερο να καταλάβουμε ποιες, ποιοι είναι οι λόγοι της ρήξης και να θελήσουμε να επανε, δημιουργήσουμε μια εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και των ανθρωπιστικών ήμουν ο στρατιωτικός υπεύθυνος εκεί των 25 περίπου στρατιωτικών οργανώσεων που συνεργάζονταν εκεί. Η εκ νέου δημιουργία των σχέσεων με τους ανθρωπιστικούς ήταν κάτι το ζωτικό. Αναθεωρήσαμε λοιπόν πλήρως τους τρόπους δράσης μας και θελήσαμε να δημιουργήσουμε νέου τύπου σχέσεις. Αποφάσισα καταρχήν να μάθω από τους υπεύθυνους των μη κυβερνητικών οργανώσεων γιατί επέκριναν τη δράση μας και είδα ποια είναι η ανθρωπιστική δραστηριότητα που πραγματοποιούσαν. Οι προσωπικές αυτές σχέσεις αναπτύχθηκαν επί 1,5 χρόνο μέσω δείπνων όπου κατάλαβα καλύτερα πώς λειτουργούσαν εκείνοι και εκείνοι πώς λειτουργούσαμε εμείς. Έτσι υπήρξε μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή στις σχέσεις μας παρά τις διαφορετικές ερμηνείες που έκανε η κάθε χώρα των στρατιωτικοπολιτικών σχέσεων. Και οι σχετικά καθαρά στρατιωτικές συναντήσεις έγιναν πιο ανθρώπινες. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα πληροφόρησης με εβδομαδιαία δελτία που ανέφερε τα ωράρια των αποστολών και τις βασικές ζώνες όπου θα δραστηριοποιούμασταν. Επίσης δεν, δεν οργανώναμε συνοδείες παρά μόνο με ρητή αίτηση της κυβέρνησης ή των ΜΚΟ. Για να μπορέσουν, ε, θελήσαμε να διευκολύνουμε την κυκλοφορία όλων, ιδίως στην εποχή των βροχών και οργανώσαμε τις πτήσεις. Οργανώσαμε εργαστήρια ευαισθητοποίησης, στα οποία μίλησα και εγώ, και συμμετέχαμε συμμετείχαν εκεί όχι μόνο οι ειδικευμένες ομάδες αλλά και οι υπεύθυνοι στρατιωτικών μονάδων και δέχτηκα 8 προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που η πρότειναν η ΜΚΟ και διήφθηνα εγώ. Τέλος, οι 10.000 Ευρωπαίοι στρατιώτες που υπηρέτησαν στο Τσάδ έμαθαν πολλά για τον τρόπο λειτουργίας των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των σχέσεων που πρέπει να δημιουργούνται για να μπορέσουν να συνδυαστούν τα στρατιωτικά με τα ανθρωπιστικά. Τώρα, το πρόγραμμα παρέμβασης για τους αμάχους της Λιβύης αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι αρχές του Όσλο και ελπίζω οι, όσοι θα αναλάβουν την επιχείρηση αυτή πράγματι να τις εφαρμόσουν με την καλή θέληση που είναι πάντοτε βέβαια απαραίτητη. Μια διευκρίνηση και μόνο. Προσπαθήσαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσκαλέσουμε και στρατιωτικούς, αλλά για λόγους καθαρά ε, ε, δικούς τους ήταν αδύνατον να έχουμε στρατιωτικούς να παρίστανται σήμερα το πρωί για λόγους προσωπικούς τους και προσωπικού προγράμματος. Η κυρία Μακδόναλντ έχει το λόγο από πλευράς προσφύγων της Νορβηγίας. Um, um Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω τους προηγούμενους ομιλητές καταρχήν και να ευχαριστήσω για την ε, πρόσκληση και την υποστήριξη στο Συμβούλιο Προσφύγων της Νορβηγίας. Είμαστε μια οργάνωση που υπάρχει 60 χρόνια. Εγώ εργάζομαι σε 20 χώρες. Πολλά από τα θέματα που ήθελα να θέσω για τις αρχές καλύφθηκαν από προηγούμενους ομιλητές, οπότε περνώ κατευθείαν στα πρακτικά θέματα. Τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν στο Αφγανιστάν, ε, ασχολήθηκα με ε, θέματα στρατητικά και πολιτικά, ήμουν πρόεδρος στην ομάδα συντονισμού και αξιοποίησα την εμπειρία από το Σουδάν όπου πήγα για να ε, ασχοληθώ πάλι με τη συνεργασία ανθρωπιστικών στρατιωτικών φορέων. Όταν πρόκειται λοιπόν για το ρόλο των αρχών, εδώ πρόκειται για θέματα αντίληψης και αποδοχής. Όταν πήγα πρόσφατα στις Φιλιππίνες και ε, πήγαμε να παρέμβομαι σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις παγκοσμίω εκεί, το όλο θέμα της αποδοχής από τους παράγοντες εκεί και η αποδοχή από την κυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν τις ε, αρχές αυτές ότι είμαστε εκεί για τις ε, ανάγκες του κόσμου και δεν ε, πήραμε θέση υπέρ ενός από τα μέρη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μας θεωρήσουν ότι δεν συνιστούμε απειλή. Είμαστε για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, όχι τις ανάγκες της μιας πλευράς. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Θα μιλήσω για τις διεθνείς ε, στρατιωτικές δυνάμεις. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον ε, αφορά το ρόλο των ε, στρατιωτικών φορέων. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για τις διεθνείς, όχι τις εθνικές, και τις συγκρούσεις. Στο Αφγανιστάν κάναμε πολλές συζητήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε τις στρατιωτικές πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίστηκαν πριν από λίγα χρόνια και επί τρία χρόνια προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές οι ενεχόμενοι εκεί. Θεωρητικά επί χάρτου είναι καλές αλλά δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη, αποτύχαμε για διάφορους λόγους. Και εδώ πάνω σε αυτό θα μιλήσω. Ένας βασικός λόγος ε, είναι το θέμα αυτό της εκστρατείας που θα πείσει ε, συναισθηματικά και εγκεφαλικά ε, υπέρ της σταθεροποίησης. Κυρίως ε, πρόκειτο για την προστασία των δυνάμεων. Πολλοί ήθελαν να το εξασφαλίσουν αυτό, κερδίζοντας τον πληθυσμό και παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό που είδαμε στο Ανατολικό Αφγανιστάν ήταν ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είχαν ε, προβλήματα γιατί στο περιβάλλον εργασίας τους οι στρατιωτικές δυνάμεις παρήχαν ιατρικές υπηρεσίες και εκείνοι, οι μη στρατιωτικοί επίση που δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες, ακολουθούσαν τις ίδιες διαδικασίες, δούλευαν για τους ίδιους ανθρώπους και πολλές φορές ε, έρχονταν ε, ε, ε, αντιστασιακοί στη χώρα και έκλειναν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μετά αποφασιζόταν να επιχειρηθεί κάτι το διαφορετικό και δεν υπήρχε ε, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα βοήθειας, δεν λειτουργούσε μακροπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε όχι μόνο τις αρχές αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Πολλοί είχαν ε, παλιά στρατιωτικοί, είχαν πρόσβαση σε ε, ιατρικές υπηρεσίες, τώρα δεν έχουν. Πολύ συχνά μας λένε ότι ε, λυπάται, ε, λυπούνται οι ένοπλες δυνάμεις στον ε, κόσμο, το λαό εκεί. Ο κόσμος έχει δικαίωμα υποστήρι, να υποστηριχθούν. Μπορεί να είναι ανάμεκτες οι ανάγκες. Εμείς είμαστε έμπειροι ε, επαγγελματίες, 60 χρόνια υπάρχει η δική μου η οργάνωση, υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά που κάνουμε. Αυτό που είδαμε στο Δυτικό Αφγανιστάν είναι ότι γινόταν διανομή ε, εξοπλισμού σε σχολεία. Ε, την επόμενη μέρα ο εξοπλισμός αυτός επολύτως στην ε, μαύρη αγορά λόγω της διαφοράς που υπάρχει. Ήταν λοιπόν κακή βοήθεια αυτή. Τυφλοί για τους οποίους προορίζονταν η βοήθεια δεν την έλαβαν και ε, όλοι ε, περίμεναν τι θα αποκόμιζαν τα διάφορα προγράμματα. Επίσης, ε, το, η επίπτωση που έχει το CNN και το BBC είναι πιο εύκολο να θεωρηθεί ότι δίνουμε μπάλες ποδοσφαίρου ή βιβλία και όλοι και οι, οι στρατιωτικοί σε σχέση με αυτό είναι σε δύσκολη θέση γιατί αυτά θέλει ο κόσμος δεν θέλει την, να δει την πραγματικότητα αναγκαστικά και εμείς ε, ε, τους πιέσαμε και τους στρατιωτικούς αν θέλετε να αναλάβουν ανθρωπιστική δράση. Όταν δουλεύουμε επί τόπου με τους στρατιωτικούς φορείς βλέπουμε να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες στη θέση τους πώς θα αντιμετωπιστούν από τον ε, ντόπιο πληθυσμό δηλαδή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, η σύγχυση των ρόλων δεν είναι ε, πάντοτε αθέλητη, καμιά φορά είναι και σκόπιμη. Ε, το είδαμε και με τα λευκά οχήματα που τα χρησιμοποιεί και ο στρατός. Ε, αυτά δεν αποτελούσαν στόχο, αυτό ήταν ο σκοπός, αν οδηγεί στο δρόμο και υπάρχουν κάποια, ε, κάποιες αντιπολιτευόμενες ομάδες ε, στο δρόμο, πώς θα καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ ημών και των στρατιωτικών. Για να είμαστε ειλικρινείς, ε, δεν είναι θεμητός στόχος οι ε, πολίτες, οι άμαχοι και οι άμαχοι θα πρέπει να προστατεύονται. Αυτό που είναι λοιπόν χρήσιμο είναι μπορούμε να επικεντρωθούμε γιατί έχουμε πολλές κατευθυντήριες γραμμές. Πώς θα εφαρμοστούν όμως όλες αυτές. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ θα είναι πολύ θετικό. Για τη σταθεροποίηση δύο λόγια. Η σταθεροποίηση ε, περιλαμβάνει πολλές ολοκληρωμένες ε, ε προσεγγίσεις. Ε, είναι θέμα ορισμού. Ε, θα πρέπει και εδώ οι στρατιωτικοί να ενταχθούν στην διαχείριση των κρίσεων. Πώς αντιμετωπίζεται η σύγκρουση, ποιοι είναι οι συγκρουόμενοι. Ε, πολλές φορές θα πρέπει να βάλουμε στην πρώτη γραμμή την προστασία των πολιτών. Οι γιατροί, οι ασθενείς, πολλές φορές γίνονται πιόνια και εργαλεία σε μια σύγκρουση. Είναι αυτή οι οποίοι μένουν εκεί αφού αποχωρήσουν οι στρατιωτικοί και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις όταν επισέλθουν άλλοι παράγοντες και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σε μία σύγκρουση, έτσι αυξάνονται για αυτούς οι κίνδυνοι. Αυτό είναι σημαντικό σε μια μεταβατική φάση που περνάμε τώρα το Αφγανιστάν. Όταν φύγουν οι στρατιωτικοί, τι θα κάνουν αυτοί που παίρνουν οι παραλήπτες της βοήθειας ή εμείς των ανθρωπιστικών οργανώσεων τι θα κάνουμε αν θεωρηθεί ότι υποστηρίξαμε τη μία πλευρά ε, στη σύγκρουση. Είναι ένα πραγματικό θέμα αυτό. Επίσης, ε, για να επανέλθω στην αντίληψη, πώς μιλάμε για τη σύγκρουση, Πολλές φορές κάνουμε δηλώσεις ε, δημόσιες ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το βλέπουμε και στη Λιβύη, όπου ένας αρχηγός κράτους είπε πρόσφατα ότι η Λιβύη είναι σε ανθρωπιστικό πόλεμο. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε επί τόπου αυτό το πράγμα, αυτή τη δήλωση, όταν δηλώνουμε ότι εμείς κάνουμε, θέλουμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια ε, και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Επίσης θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός είναι σημαντικός, η ότσα παίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό ε, πολιτικών στρατιωτικών φορέων ε, σε ένα περιβάλλον σύγκρουσης. Η ΕΚΟ επίσης είναι πολύ σημαντική ε, επιτόπου ως δωρητή και έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί πρωτίστω βάσει αρχών. Αυτό είναι κάτι που το εκτιμούμε πολύ. Νομίζω ότι τέλειωσε ο χρόνο μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Nous allons... Euh, ευχαριστώ πολύ. Αρχίζουμε με τις ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σούλα. Pardon. Je me disais bien, je ne connais pas son nom, mais monsieur à ma droite écrit très mal. Ε, δυστυχώς, ο γραφικός σας χαρακτήρας δεν είναι και πολύ καλός. Ο κύριος Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η πληροφόρηση ήταν καλή. Πριν από χρόνια είχαμε επισκεφθεί το Κονγκό στα πλαίσια της συνέλευσης ΑΚΕ ε, Ένωσης και πρέπει να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε τότε πολύ και από τις ε, εξελίξεις και από την ε, κυβέρνηση Καμπίλα. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες τότε. Δεν είχαμε την εντύπωση ότι θα υπήρχε με τους αντάρτες ε, σύγκρουση. Εσείς τώρα μας τα είπατε διαφορετικά, οπότε υπάρχουν εδώ κάποιες εξελίξεις που οδηγούν σε ανησυχίες σε σχέση με ενδεχόμενο πολεμικών συγκρούσεων. Σε σχέση με τις εκλογές τι γίνεται. Θα γίνουν κανονικά, νομότυπα οι εκλογές. Ο πρόεδρος στην Ανατολική χώρα πήρε πολλές ψήφους. Τι γίνεται με τον μόνιμο αντίπαλό του όποιος έχασε παρατρίχα τις εκλογές αλλά εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ως πολιτικό πρόσωπο στη διαδικασία των εκλογών τι αντιπαράθεση θα γίνει. Στην Ανατολή οι αντάρτες μπορεί να αυξήσουν τη δύναμή τους και αυτό πάλι να οδηγήσει σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Αυτό θα ήταν πολύ ανησυχητικό. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να απαντήσετε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ε, άλλες έτσι. Α, ο κύριος ε, Γκέρενς. Ο κύριος Γκέρενς. Όχι, δεν έγραψε ο διπλανός σας ε, γιατί δεν είχα δηλώσει το όνομά μου. Ως προς το Αφγανιστάν, Αναζητούμε τους ε, πραγματικούς λόγους ε, για τους οποίους μπορεί να πληγεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Καταρχήν η ανθρωπιστική βοήθεια εξεδίωξε τους Ταλιμπάν ή τουλάχιστον ε, μείωσε την επιρροή τους μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μετά είχαμε και του στρατιωτικούς που είχαν καθαρά ένα ειρηνευτικό έργο. Μετά όμως είδαμε ότι υπήρξαν πραγματικοί κίνδυνοι έναντι των υπευθύνων της ανθρωπιστικής βοήθειας και πολλές φορές δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ ε, στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους. Υπάρχουν μη κυβερνητικέ οι οποίες αρνούνται οποιαδήποτε συγχρηματοδότηση εάν η χώρα τους συμμετέχει σε μια πολεμική σύνεργα. Ξέρω για μια μη κυβερνητική η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε συγχρηματοδότηση τη στιγμή που υπήρχαν άλλες χώρες που συμμετείχαν στην, στις πολεμικές επιχειρήσεις του Κόσοβο. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο τη στιγμή που αποκόπτεται κάθε δεσμός, κάθε σύνδεσμος, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά ίσως τις υποβάλω αργότερα. Και εγώ έχω μία ερώτηση, υπάρχει άλλη μία ερώτηση από την κυρία Τζίμερ. Ο μιλητής μας ε, είπε για την ανθρωπιστική δουλειά από στρατιωτικούς φορείς είπε ότι είναι μια μακρά διαδικασία όπου οι στρατιωτικοί, οι ένοπλες δυνάμεις έμαθαν πολλά πράγματα για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δεν είναι μακάβριο να υποθέτουμε ότι τέτοιε εμπόλεμε ζώνες και περιοχές, σε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γίνονται, αν θέλετε, ε, ευκαιρίες για να μάθει ο στρατός, όπως λέμε στο κασίδι το κεφάλι. Ε, έτσι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και οι στρατιωτικοί οι οποίοι ε, μετά από πολεμικές επιχειρήσεις ε, υφίστανται ψυχολογικά τραύματα και άλλα προβλήματα και μετά περνούν, στην καλούνται να συμμετάσχουν στην ανθρωπιστική ε, βοήθεια με αποτέλεσμα πολλοί να στρέφονται, από τον τόπιο πληθυσμό να στρέφονται εναντίον τους Πώς θα μπορούν λοιπόν με αξιόπιστο τρόπο να παρέχουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω αυτό. Δεν αρκεί να πούμε ότι έχουμε μια μακρά διαδικασία μάθησης αν θέλετε σε αυτό το τομέα. Και επιτόπου πώς το αντιμετωπίσατε. Μήπως δηλαδή είναι μια αυταπάτη αυτό το πράγμα ότι μπορεί να γίνει. Ο κύριος Νέλχαρτερ. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο λίγες οι ερωτήσεις γιατί θα κάνω άλλη μία. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μας είπε η κυρία Μακδόναλντ και μου κάνει εντύπωση ότι μίλησε πιο πολύ για τη σύγκρουση μεταξύ των ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων παρά την σύνδεση μεταξύ τους για την παροχή βοήθειας. Εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ με την κυρία Τσίμερ γιατί στο Αφγανιστάν υπάρχει σαφώς η τάση ότι μια πλευρά πρέπει να πολεμηθεί, να καταπολεμηθεί για το καλό της κοινότητας. Και μετά θα υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια και άλλες μορφές βοήθειας. Αυτά ε, ε, είναι αυτονόητα μετά, δεν ξέρω η κυρία Μακδόναλτ πώς το βλέπει που έχει πει από πολλές χώρες. Υπάρχει μια συνεχής εναλλαγή μεταξύ πολεμικών επιχειρήσεων και παροχής βοήθειας από τις αρμόδιες οργανώσεις. Όμως είδα ότι υπάρχουν περισσότερες συγκρούσεις, έτσι κατάλαβα από αυτά που είπατε, παρά συνεργασίες. Θα ήθελα, θα μια διευκρίνηση. Θα περάσουμε στις απαντήσεις. Η κυρία Μακδόναλτ θέλει να αρχίσει. Ναι, να μιλήσω για την ασφάλεια των ε, εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και για τη χρηματοδότηση. Είναι περίπλοκο το θέμα. Παράλληλα όμως είναι και αρκετά απλό όταν ε, ήμουν στο Πακιστάν. υπήρχαν ε, χρηματοδότες, διάφοροι υπήρχαν. και ορισμένοι αποκλεισμοί. Δηλαδή, ορισμένοι δωρητές αποκλείονταν από τον τόπιο πληθυσμό. Στο, στο Αφγανιστάν ε, ήταν πιο απλά τα πράγματα. Δηλαδή θεωρήθηκε η συμβολή ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων ε, ως βοήθεια ε, κατά των ε, εξεγερμένων. Μπορούσε κανείς να πάρει χρηματοδότηση από ένα δωρητή, αλλά αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα αρκεί να στηρίζονταν στο δικό μας πρόγραμμα. Μπορούσαμε έτσι να δικαιολογήσουμε την χρηματοδότηση και στον τόπιο πληθυσμό και στους άλλους εμπολέμους. Έτσι γίνεται, έτσι διαχειριζόμαστε αν θέλετε ε, τα θέματά μας αλλά και έτσι προσεγγίζουμε το θέμα της αντίληψης για το ρόλο μας από τον τόπιο πληθυσμό. Ε, στην περίπτωση του KPK έπρεπε να κάνουμε μια ανάλυση ε, και για την διαχείριση της ασφάλειας. Επίσης η ανεξάρτητη χρηματοδότηση είναι ουσιώδης εν πάση περιπτώσει. Τα κονδύλια από την ΕΚΟ θεωρούνται ουδέτερα κονδύλια, θεωρούνται ε, ανεξάρτητη πηγή χρηματοδότησης και αυτό ήταν σημαντικό. Τώρα, για την διαδικασία μάθησης θα απαντήσει και ο συνάδελφος. Εγώ να πω μόνο ότι αν δούμε το Αφγανιστάν Έχουμε 100.000 ε, στρατό, ε, διαφορετικές οργανώσεις, πολλές γλώσσες, ε, εναλλασσόμενα προγράμματα, εναλλάσσονται δηλαδή οι υπεύθυνοι. Τι διαδικασία μάθησης να υπάρχει εκεί. Εμείς είμαστε... Ε, ε, ε, η, τεχνογνωσία βρίσκεται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχει πολλούς ειδικού επαγγελματίες. Εμείς διασφαλίζουμε το πώς θα συνεχίσουμε για να καλύπτουμε τις ανάγκες, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών, των αμάχων. Τώρα, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας σχετικά με τις εμπειρίες ε, για τις ε, συγκρούσεις μεταξύ ανθρωπιστικών στρατιωτικών φορέων. Υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει και απογοήτευση. Ε, καμιά φορά οι φορείς αυτοί συνεννοούνται καλύτερα γιατί αναγνωρίζουν ότι ο στρατιωτικοί, οι στρατιωτικοί είναι για να αντιμετωπίσουν τη σύγκρουση, οι ανθρωπιστικοί φορείς απαλύνουν τα δεινά των στρατιωτικών συγκρούσεων. Ε, παρεμβαίνουν οι πολιτικοί και προσπαθούν να διακινήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια. Αυτό είναι το προτιμητέο και όχι να συμβάλλουμε σε μια σύγχυση. Δεν... Μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Οι πολιτικές στρατηγικές καμιά φορά δημιουργούν σύγχυση των ε, ρόλων και των ταυτοτήτων. Καμιά φορά για λόγους δικούς τους. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο δεν ετέθη ως προς το στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος συνεργασία. Θα ήθελα να είμαι κάπως προκλητικός. Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης ε, μεταξύ στρατιωτικών και υπευθύνων ανθρωπιστικής βοήθειας στο Τσάντ. Ε, δηλαδή είναι μια ιστορία αγάπης, άρχισε πολύ καλά, προχώρησε μέτρια και δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει για να απαντήσω πιο σοβαρά στο ερώτημα που ετέθη από την κυρία Τζίμερ για την κατάρτιση. Δεν υπάρχει εμφυσιμία σε αυτό που είπα. Δηλαδή 10.000 στρατιωτικοί κάτι έμαθαν. Ήμασταν εκεί όμως για να, κάνουμε, για να επιτελέσουμε ένα έργο. Δεν πήγαμε για να μάθουμε κάτι καινούριο, μία νέα ε, τεχνογνωσία. Αυτό Ελπίζω να το αποδείξαμε, αλλά υπήρξε ένα άνοιγμα αυτών των στρατιωτών και των αξιωματικών, ένα άνοιγμα προς ένα νέο κόσμο. Και έμαθαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαζε τα σήματα από τα οχήματα και έπρεπε να τους εξηγήσουμε ότι αυτό είχε λόγο, λανθασμένα ή όχι. Τους εξέπληξε το γεγονός ότι δεν έπρεπε να κάνουν σχέδια για τους πληθυσμούς, γιατί πολλές φορές οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ήταν απασχολημένες αλλού, σε άλλους καταβλισμούς προσφύγουν. Έπρεπε να να βοηθήσουν τους πληθυσμούς εκεί που το ζητούσα εγώ. Δεν ήταν εύκολο για αυτούς που είχαν πείρα στο Αφγανιστάν. Το Force Protection που αναφέρεται δεν έκανε προβολές έργου υπέρ των πληθυσμών, αλλά έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα. Και για αυτούς δεν ήταν εύκολο να κατανοήσουν ότι μιλάμε για 60 φυλές διαφορετικές που μιλούν και διαφορετική γλώσσα. Το μάθαν βαθμία μαθαίνοντας τον πολιτισμό. Γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε με την εκστρατεία Hearts and Mind για να το μάθουν αυτό. Πρόκειται για ένα άνοιγμα ε, προς ε, τους υπεύθυνους ανθρωπιστικής βοήθειας και ελπίζω οι στρατιωτικοί να το ε, χρησιμοποιήσουν καλύτερα στο μέλλον. Υποστηρίξτε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες έτσι ώστε οι χώρες που εκπροσωπείτε να μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες. Εργάζομαι του θέματος, υπάρχει μεγάλη τεκμηρίωση αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα προσέγγισης γιατί είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Ήρθα σε επαφή με τις στρατιωτικές δυνάμεις των Μένων Εθνών και ξέρω ότι είναι δύσκολο να υποστηριχτεί κάτι τέτοιο. Είναι, πρέπει να βοηθήσουμε αλλήλους έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να επιτελέσει το έργο του. Ο Καμπάμπα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Υπάρχει μία αρνητική προσέγγιση γιατί υπάρχει αρνητική εξέλιξη. Μετά το 2006, μετά τις εκλογές, είχαμε πολλές πολιτοφυλακές οι οποίες δεν ελέγχονται στο ανατολικό μέτωπο του Κονγκό. Σε όλο το ανατολικό μέτωπο από βορρά προς νότο. Και αυτές οι ομάδες είναι δραστήριες, τροφοδοτούνται από την λαιλασία φυσικών πόρων και στο ανατολικό αυτό μέτωπο επίσης του Κονγκό οι στρατιωτικοί και οι κιανόκρανοι προσπαθούν να προστατεύσουν ε, τους πολίτες. Αυτοί οι 8.000 κιανόκρανοι δεν μπορούν να δράσουν. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή είτε έχουμε σωρία κιανόκρανων που δεν μπορούν να προστατεύσουν τους ε, ε, πολίτες και από την άλλη πλευρά έχουμε δυσκολία να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς που έχουν ε, πληγεί. Υπάρχουν και ντόπιοι αντάρτες, αλλά και ξένες ομάδες από το Μπουρούντι, από τη Ρουάντα, από το, την Ουγκάντα και από το Σουδάν, που βρίσκονται στο ανατολικό μέτωπο του Κονγκό και είναι δύσκολο να παρέμβουμε διότι υπάρχουν μεγάλοι κλειδονισμοί στο ανατολικό μέτωπο και οι άμαχοι αναρωτιούνται τι θα γίνει. Ως προς εκλογές θα ήθελα να πω ότι και πάλι θα πρέπει να ορίσουμε ποιοι είναι οι ψηφοφόροι, να γραφτούν στους εκλογικούς καταλόγους και με όλους αυτούς τους καταβλισμούς είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η καταγραφή. Ως προς τις εκλογές υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι πολύ δύσκολο η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό να διοργανώσει τις μελλοντικές εκλογές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η προστασία τις εκλογικής διαδικασίας. Υπάρχουν διάφορες, διάφορα αντάρτικα που είναι δραστήρια στο Κονγκό και μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Επίσης υπάρχει αποδυνάμωση των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως έχουμε συμμετοχή 20.000 ατόμων αλλά υπάρχει αποδυνάμωση αυτών των ε, δυνάμεων. Επίσης, η ανεξάρτητη οργάνωση διενέργειας εκλογών δεν ε, μπόρεσε να αναλάβει δράση. Και έναντι όλων αυτών των ε, δυσκολιών θα γίνει αναβολή των εκλογών ίσως διενεργηθούν το 2012. Ως προς την άλλη σας ερώτηση για τις προβλέψεις και την προεκλογική εκστρατεία, είναι δύσκολο να περάσουμε από δύο γύρους σε έναν και ο απερχόμενος υποψήφιος ε, είναι σε καλύτερη θέση, ε, διότι οι ψηφοφόροι ψηφίζουν για τον ε, υποψήφιο της περιφέρειάς τους, όχι για μίας άλλης. Άρα, επειδή έχει μεγαλύτερο πληθυσμό το ανατολικό μέτωπο, το ανατολικό Κόγκο, ίσως σε αυτή την περίπτωση υπάρξουν δυσκολίες. Το 2006 εξελέγει διότι μίλησε υπέρ της ειρήνης. Ο, το ανατολικό μέτωπο, στο ανατολικό μέτωπο δεν υπάρχει ειρήνη. Άρα, ο Ζαν Πιέρ Μπέμπα θα του δημιουργήσει δυσκολίες διότι θα δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπάρχει ο Ετιέν Σεκεντή, ο οποίος είχε αντιταχθεί στο όμομπό του και ο οποίος δεν είναι ούτε από την Ανατολή ούτε από τη Δύση. Το κέντρο του Κονγκό δεν έχει τόσο υψηλό, τόσο μεγάλο πληθυσμό. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αντιρρήσεις και ίσως λάβει αρκετές ψήφους α, με μαθηματική ακρίβεια. Μπορώ να πω όμως ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο Ετιέν Σεκεντή μάλλον δεν θα κερδίσει αυτές τις ε, εκλογές. Γκέρενς, άλλη μια ερώτηση πριν περάσουμε στο τρίτο πάνελ που είναι και το τελευταίο. Ως προς το στρατιωτικό και το πολιτικό σκέλος. Εάν, ε, το ε, οι στρατιωτικοί επιτελούν και το ανθρωπιστικό έργο, τότε είναι ένστολοι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που δεν είναι ένστολοι. Άρα, επειδή μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθαρά, ε, οι μεν δεν εντάσσονται στους δε. Δηλαδή υπάρχουν οι ένστολοι και οι μη ένστολοι που διατρέχουν κίνδυνο. Εσείς είπατε ότι η ΕΚΟ θεωρείται ένα ουδέτερο μέτωπο. Άρα οι αξιωματούχοι της ΕΚΟ δεν διατρέχουν κινδύνους, τόσους κινδύνους. Άρα οι υπεύθυνοι ανθρωπιστικής βοήθειας βρίσκονται επιτοπίως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενώ εκείνοι που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια παραμένουν για μεγάλες χρονικές περιόδους. Δεν χρηματοδοτούνται όμως από τις ίδιες πηγές. Άρα, για να υπάρχει ασφάλεια και των μεν και των δε, δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ΕΙΕΔ που αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη πολιτικής δράσης και να τη διαχωρίσουμε από την ίδια την αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των ε, δύο σκελών. Ξαναθέτω το ερώτημα γιατί η Λέδη Άστον δεν είναι σαφής επί του θέματος. Τι θα συμβεί όταν το αναπτυξιακό σκέλος έρθει σε ρήξη με ένα άλλο σκέλος που είναι το στρατιωτικό. Πώς θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα. Δεν είσαστε της άποψης ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να τεθεί κάνοντας διάκριση μεταξύ ΕΙΕΔ και αυτής της διάστασης, διότι αν εάν αφήσουμε το ανθρωπιστικό σκέλος τότε ε, δηλαδή το ε, ανθρωπιστικό σκέλος καθαρά ως προς την επιμελητιακή βοήθεια δεν θα τα καταφέρουμε καθόλου καλά. Διότι αυτός είναι ο απότερος στόχος, η ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Μπορεί κάποιος να απαντήσει. Ο κύριος Καμάμπα, σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να δούμε πώς ορίζουμε την αποστολή. Όταν μιλάμε για στρατιωτική δράση, η στρατιωτική δράση δεν ορίζεται επακριβώς. Υπάρχει ένα μέρος που ορίζεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά στη θέση σε εφαρμογή μπορεί να υπάρξει σύγχυση. θα μπορούσαμε να έχουμε μία καταπροσέγγιση ανάλυση της επιτόπιας κατάστασης. Μιλώντας για στρατιωτική δράση, γιατί θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα και έτσι θα προωθήσουμε τη βοήθεια, τότε μόνο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πληγέντες. ο ρόλος των στρατιωτικών δεν είναι σαφής και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έχει τεθεί η συζήτηση και για τους κιανόκρανους όπου μιλάμε για την τρίτη γενναία κιανόκρανων οι οποίοι θα είναι πολυλειτουργικοί. Μπορούν να προστατεύσουν τους πληθυσμούς, είναι εμπόλεμοι, μπορούν να χτίσουν γέφυρες και ούτω καθεξής. Και από, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα μπορέσει κανείς να διαφύγει από αυτή την ε, εικόνα σε αδρές γραμμές εάν δεν ορίσει ακριβώ τις αποστολές με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο. Διότι in του βλέπουμε ότι πολλές φορές αλλάζει η αποστολή χωρίς να, αλλάζει το κείμενο. Κύριε Μακδόναλντ. Um, Νομίζω ότι πως ε, πρέπει να είναι χωριστή η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό θεωρούν πολλές οργανώσεις. Η πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής έχει πρακτικές επιπτώσεις, όπως το Αφγανιστάν που φαίνεται. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αμφισβητούν τη συνεργασία ακόμα και με τον ΟΗΕ μετά από δυσάρεστες εντυπώσεις. Γιατί και εκεί και ο ΟΗΕ είναι πολιτικοποιημένος. Θα ήταν τραγικό να συμβεί το ίδιο και με την ΕΚΟ που είναι τόσο σημαντικός ανθρωπιστικός δωρητής, χρειάζεται προσοχή να μην ε, πολιτικοποιήσουμε την ανάπτυξη, γιατί αυτό, ε, ας πούμε, στο Αφγανιστάν οι στρατιωτικοί μπορεί να ε, λένε ότι οι σκηνές τα τρόφιμα, οι κουβέρτες είναι ανθρωπιστική βοήθεια και όλα τα άλλα είναι αναπτυξιακή. Όταν αντιμετωπίζουμε με κατεπίγουσα ανάγκη θα πρέπει ο πολιτικός τομέας, ο μη στρατιωτικός να διαχωρίζεται από τον στρατιωτικό. Ε, οπωσδήποτε η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να διαχωρίζεται, αλλά και η ανάπτυξη στηρίζεται στις ε, ανάγκες και δεν πρέπει να ε, κυριαρχείται από τους στρατιωτικούς. Καλό θα είναι να μην στρατιωτικοποιείται και πολιτικοποιείται η βοήθεια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω, αν και άμεσα δεν μπορώ γιατί δεν έχω τις ικανότητες. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να τονίσω κάτι σημαντικό που λέγεται στις Ηνωμένε Πολιτείε Stabilization Industry. Δηλαδή, αυτούς που βλέπετε με στολή αυτή τη στιγμή αλλά που αύριο θα είναι χωρίς στολή με πολιτικά και θα έχουν άλλες αρχές εφαρμογής από αυτές που εφαρμόζουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Υπάρχει πάντως μία σύνδεση, διότι αυτή η βιομηχανία της σταθεροποίησης έχει ξεπεράσει το στάδιο της άμεσης ε, πήγουσας κατάστασης και της χορήγησης βοήθειας και τώρα χορηγεί υπηρεσίες ασφαλείας, μεταφορών, εξυγίανσης κλπ. Και τώρα ασχολούνται και με θέματα ανάπτυξης. Πρέπει να περάσουμε στην τρίτη συζήτηση. Μήπως θέλετε να θέσετε το ερωτήματά σας μετά, μετά, γιατί όλα συνδέονται. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί. Το πολιτικό πρόβλημα σε εμά τίθεται. Το θέμα δεν είναι απλώς να προασπίσουμε τους ανθρωπιστικούς που πρέπει, αλλά και εκείνου που παραμένουν επί τόπου πιο μακροχρόνια και διατρέχουν ακριβώς τους ίδιους κινδύνους. Αντίθετα, εάν θέλουμε η εικόνα είναι ουδέτερη, τότε πρέπει και οι πηγές χρηματοδότησης που τροφοδοτούν όλες αυτές τις επιχειρήσεις να είναι και αυτές ουδέτερες και τότε πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα ως προς την διοργάνωση της λειτουργίας της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Συμφωνώ απόλυτα κύριε Γκόρεντς. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην τρίτη συζήτηση γιατί η δεύτερη τελείωσε. Λοιπόν, ο κύριος Μαρτέν Λακούρ είναι εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων στο αρχηγείο Ερυθρού Σταυρού των Βρυξελών και την κυρία Καρίμα Φαρίμη που είναι της Oxfam. Α, δεν ευχαρίστησα τους προηγούμενους ομιλητές και ομιλήτριες. Θα αρχίσουμε τώρα για να μην χάνουμε χρόνο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαρτίνο Λακούρ. Έχετε και διαφάνειες, α, μάλιστα. Next for the one the Right. Um, hello. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να σας συναντήσουμε. Φοβάμαι ότι πολλά πράγματα αναγκαστικά θα τα επαναλάβω. Όμως πολλές φορές η επανάληψη δεν είναι τόσο κακό πράγμα. Θα αρχίσω σε πρακτικό επίπεδο, στο επίπεδο του πεδίου της μάχης. Και αν κάποιος παρακολουθεί τους ανθρωπιστικούς και τους στρατιωτικούς φορείς, θα παρακολουθεί και τη πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Αφγανιστάν πριν από λίγα χρόνια. Αυτά είχαν υποθεί που βλέπετε στο, στη διαφάνεια. Υπάρχουν σε αυτή τη δήλωση τέσσερα βασικά μηνύματα. Πρώτον, η εγκύτητα και η ευελιξία των ανθρωπιστικών φορέων που αναγνωρίζεται από κάποιον που θεωρεί το 20 χρόνια πριν από όλα τα έθνη ως αγωνιστής για την ελευθερία. Ενώ τώρα θεωρείται εξτρεμιστής ή και τρομοκράτης. Η εγκύτητα, η ευελιξία λοιπόν αναγνωρίζεται. Η ουδέτερη δράση μπορεί να επενείται ακόμα και σε πολύ πολλωμένο περιβάλλον όπως το Αφγανιστάν. Η πολιτιστική περιχαράκωση μπορεί να ξεπεραστεί. Όχι να ε, πληρωθούν τα κενά, αλλά μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να παρουσιαζόταν ε, αυτές οι δηλώσεις ως δυτικές. Αναμφίβολα γνωρίζει ο, αυτός που τα λέει αυτά τις πηγές της χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά η ουδέτερη δράση του επιτρέπει να, επιτρέπει να γίνει αποδεκτή η δράση του Ερυθρού Σταυρού στο Αφγανιστάν. Αυτή ήταν μια πρακτική δήλωση που έγινε επί τόπου. Ένα μια δήλωση από έναν επικεφαλής ε, Ταλιμπάν που θα ε, ανατραπεί από μια δήλωση του Anders Fogg Rasmussen στο Σικάγο το 2010. Πάλι υπάρχει ένα ενοιολογικό θεωρητικό θέμα εδώ, φεύγουν από το πεδίο της μάχης. Βλέπουμε όμως, και αυτά που θα σας πω ήδη υπογραμμίστηκαν και προηγουμένως σήμερα το πρωί. Υπάρχουν όμως δύο ε, βασικές παρανοήσεις. Πρώτον, ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα, σε κάποια δεδομένα πλαίσια, ενώ αυτό δεν αληθεύει. Αν, αν πούμε ότι είμαστε στο ίδιο ποτάμι, εντάξει, αλλά στην ίδια βάρκα δεν είμαστε. Και να μιλήσω τώρα για τους στρατιωτικούς. Εκείνοι ίσως έχουν σκάφη ε, δυνατά. Ως επιτοπλίστων οι ανθρωπιστικοί φορείς ε, έχουν πιο μικρά ε, πλοία αλλά ξέρουν το ποτάμι όπως αναγνωρίστηκε και από τον αρχηγό των Ταλιμπάν. Οι ανθρωπιστικοί ως επιτοπλίστων ζουν για κάποια χρόνια σε μια περιοχή ή δεκάδες χρόνια. Αυτή η παρανόηση ότι είναι στην ίδια βάρκα όλοι προέρχεται από το ότι συμμεριζόμαστε το ίδιο πολιτιστικό υπόβαθρο, η στρατιωτική και η ανθρωπιστική. Οι Γάλλοι στρατιωτικοί καμιά φορά δυσκολεύονται να καταλάβουν έναν αντιπρόσωπο Ελβετό από τον ε, Ερυθρό Σταυρό που δεν συμμερίζεται καμιά φορά τις ίδιες ε, αξίες. Το ίδιο ισχύει και για την ουδετερότητα. Και εκεί νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας Ράσμουσεν λέει ότι για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ε, μια ιερή αρχή η ουδετερότητα και ότι δίνονται μάχες αρχών χωρίς να γίνεται κατανοητό ότι η ουδετερότητα είναι μόνο ένα μέσον που εξυπηρετεί ένα σκοπό είναι η δική μας πανοπλία, είναι το επιχειρησιακό μας εργαλείο. Αυτή η διαφάνεια επαναλαμβάνει το ίδιο ότι δεν είναι όλοι οι φορείς που συμμερίζονται τους ίδιους στόχους. Ίσως στη δεύτερη παύλα πρέπει να προσθέσω ότι αν οι ανθρωπιστικοί, φο... ανθρωπιστικοί φορείς δεν ε, φροντίζουν ε, είναι, δεν είναι κράτη. Αν ήταν τότε θα υπήρχαν και θα είχαν δράσει και στην Κολομβία και στη Σομαλία και οπουδήποτε υπάρχουν ανθρωπιστικές ανάγκες. Το γεγονός ότι γίνεται επιλογή που θα παρέμβουν τα κράτη σημαίνει ότι δεν είναι ανθρωπιστικοί φορείς. Ακόμα κι αν συμβάλλουν στην ανθρωπιστική δράση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Για την ουδετερότητα πάλι είναι μια συμπεριφορά, μια προσωπική συμπεριφορά, μια θεσμική συμπεριφορά και καθίσταται ορατή μόνο εν δράση. Αλλιώς δεν σημαίνει απολύτως τίποτε. Επόμενο. Πολύ γρήγορα θα το προσπεράσουμε αυτό το θέμα γιατί τα έχουμε πει όλα ήδη. Περιορίζομαι μόνο να πω ότι ε, σε τελευταία ανάλυση η διαφορά δεν είναι δεν συνίσταται στην ομοιομορφία ή στην έλλειψη της ομοιομορφία ή η διαφορά δεν συνίσταται στο αν υπάρχουν όπλα ή όχι. Η διαφορά βέβαια είναι μεταξύ πολιτικής δράσης που δεν είναι κακιά λέξη και της ανθρωπιστικής δράσης. Αυτό κάνει τη διαφορά. Η συζήτηση με, ε, για τη διαφοροποίηση, συντονισμό ας πούμε, πολιτικών, στρατιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα κομμάτι ευρύτερη συζήτησης ε, που αφορά τη διαφορά μεταξύ πολιτικών, στρατιωτικών δράσεων τη μια και ανθρωπιστικών από την άλλη. Τώρα, ε, οι σχέσεις ε, πολιτικών, στρατιωτικών ο Διεθνής, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ποτέ δεν ε, φοβήθηκε το, του, στρατιωτικού. στρατιωτικούς το Ερυθρό Σταυρό το κίνημα αυτά παιδεία της, των μαχών. Και αν η καθημερινή δουλειά κάποιου είναι στο πεδίο της μάχης, ε, δεν γίνεται να αποφύγει κανείς τις σχέσεις με τους στρατιωτικούς, είτε πρόκειται για ε, κρατικούς φορείς, μη κρατικούς, αστυνομίες κλπ. Δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί η εντολή του Ερυθρού Σταυρού χωρίς να συνεργάζονται. Είναι... Και αφού ε, λειτουργούν στον ίδιο χώρο πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τους στρατιωτικούς της ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως ε, θα πρέπει να εξαρτώνται και για την ασφάλεια από αυτούς. Μιλάμε για θέματα ασφαλείας στη Λιβύη. Πάντοτε πρέπει να εξηγούμε ότι όταν μιλάμε για ασφάλεια σε σχέση με το στρα... τους στρατιωτικούς δεν ζητάμε προστασία από αυτούς. Εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρχει συντονισμός κινήσεων ε, σε σχέση και με τις ε, δυνατότητες που έχουμε και το, τις ε, δικές μας ευκολίες ούτω ώστε να έχουμε σωστές πληροφορίες κοινέ για την ασφάλεια Επίσης οι στρατιωτικές επιχειρήσεις γενικά ενεργοποιούν τις ανθρωπιστικές του, Εθνή, του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε εκτοπισμένους, ε, πληγωμένους, ε, έχουμε ε, χμαλώτους πολέμου, έχουμε κρατουμένους και θα πρέπει να συντονίζουμε τις δράσεις μας, να έχουμε διάλογο με τις αρμόδιες αρχές για να γίνονται οι δράσεις οι δικές μας. Πριν από τρία χρόνια ήμουνα στην, στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στο αεροδρόμιο είχα πάει και είμαστε τρεις σε ένα λευκό αυτοκίνητο με, που έγραφε σταυρό Σταυρός πάνω και είχαμε και ένα τέταρτο που ήταν νεκρός, που θα έπρεπε να αποδώσει στην οικογένειά του τη ο Ερυθρός Σταυρός. Κανείς από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ δεν θα πήγαινε στο χωριό για να παραδώσει ένα νεκρό. Η οικογένεια του προσώπου αυτού ποτέ δεν θα μπορούσε να έρθει στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ για να παραλάβει το συγγενή, το νεκρό συγγενή. Άρα λοιπόν, κάποιος από την ISAF θα έπρεπε να καλέσει τον Ερυθρό Σταυρό, για να αναλυφθεί αυτή η ανθρωπιστική δράση, πολύ συγκεκριμένη έστω και μικρή, χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ μας. Κάποιος από το αρχηγείο ε, ευαισθητοποιήθηκε στο τι μπορεί να κάνει ο Ερθρός Σταυρός και θεώρησε ότι η ουδετερότητα, η ανεξαρτησία, η αμεροληψία λειτουργούν και καμιά φορά είναι η μοναδική λύση. Όπως στη Λιβύη σήμερα ο Ερυθρό Σταυρό είναι ο μόνος που είναι στη Μισράτα, στη Βενγκάζη, τώρα στην Τρίπολη. Δηλαδή αυτό έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας κατευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γεράρδο, Διευθυντή του Γραφείου Σύνδεσης Βρυξελών. Ευχαριστώ κύριε Στρόφλε για το ενδιαφέρον που δείχνετε όλοι για το θέμα που και εμάς μας ενδιαφέρει. Αναρωτιόμουν αν από αυτά που άκουσα δεν θα έπρεπε να διευρύνουμε λίγο τον τίτλο της ε, ακρόασής μας γιατί νομίζω ότι μετά από αυτά που είπε ο στρατηγός φαίνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ ανθρωπιστικών δράσεων και στρατιωτικών τιάφτων έχουν βελτιωθεί. Εμείς ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το γιατί ως υπηρεσία του ΟΗΕ θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε μια τέτοια επιχείρηση κάνουν, παίζουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν. Δεν νομίζω ότι μας είδανε ποτέ ως δογματικούς. Απλώς έχουμε αρχές και θέλουμε να εφαρμόζονται. Το θέμα δεν είναι γιατί υπάρχουν αυτές οι αρχές, διότι οι αρχές αυτές δεν είναι χθεσινές και έχουν αποδειχθεί σωστές. Όπως είπε και ο Ρος το πρωί, και είναι ζωτικό το θέμα, πρέπει να δούμε πώς να προστατεύσουμε τον ανθρωπιστικό χώρο από την πολιτικοποίηση. Για μας, Είναι ιδιαίτερα σημαντικές όσο Γραφείο Βρυξελών οι σχέσεις μας με το, και με τον ΝΑΤΟ και με την Ένωση. Και η επιτυχία των σχέσεών μας με την Ένωση, στρατιωτική και πολιτική, συνίστατο στη δημιουργία ορισμένων φραγμών ή firewalls, κατευθυντήριες γραμμές δηλαδή, που να μην μπορούν, ε, που να αποτελούν όρια τι δεν μπορεί να επιβληθεί από μία κοινότητα στην άλλη. Το θέμα δεν είναι να πούμε ειδού οι κατευθυντήριε γραμμές και θα κάνετε ό,τι λένε. Είναι, το θέμα είναι ότι το στρατιωτι, η στρατιωτικοπολιτική αμυντική πόρη απαιτούν κάποιο είδους διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών για να είμαστε απλώς βέβαιοι ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα ότι δεν θα καταλήξουμε σε διαφορετική κατανόηση και σε παρεξήγηση. Οι σχέσεις λοιπόν μεταξύ ανθρωπιστικών και πολιτικών είναι κάτι που πρέπει να γίνει πιο κατανοητό. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις ο Ερυθρός Σταυρός, άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η υπηρεσία μας του ΟΗΕ συνεργάζονται με σημαντικούς παράγοντες όπως τη Σουηδία και την Βρετανία. Ο καθένας έχει ένα ρόλο να παίξει για να διατηρηθεί ο ανθρωπιστικός χώρος. Επίσης θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ήδη στην Ένωση, χάρη κυρίως στη δουλειά σας κυρία Πρόεδρε και αυτά που συζητήθηκαν στη Σύνοδο του Ιανουαρίου. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Σώμα εγκρίνει την ιδέα της ανεξαρτησίας και των άλλων αρχών που ζητάμε και εμείς. Η συνένεση των Ευρωβουλευτών για να υπάρξει αυτή η συμφωνία δείχνει τη σημασία που τις δίνουν. Όχι μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ο κοινό ορισμός της δραστηριότητας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης δείχνει. Σήμερα θα ήθελα απλώς να τονίσω τι έχει επιτευχθεί με παράδειγμα την Λιβύη. Ως υπόδειγμα παράδειγμα σχέσης. Η ανθρωπιστική κοινότητα και ο πολιτικός κόσμος και το πώς συνδυάζονται καθώς και το πώς καταλαβαίνει ο στρατιωτικός κόσμος ποιος είναι ο ρόλος του είναι το κύριο θέμα μας. Um, uh, Η... Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να δεχτεί όχι μόνο τις ανθρωπιστικές αρχές αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ε, τις εφαρμόζουν. Και αυτό πρέπει να το δεχτούν και οι στρατιωτικοί. Πολύ ενδιαφέρουσα εξελίξη είναι αυτή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι η βάση της σχέσης μεταξύ ανθρωπιστικού, πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους. Αν το ανθρωπιστικό δράση ανεξάρτητα, παρόλα αυτά πρέπει να πληροφορεί για τη δράση του τα δύο υπόλοιπα και η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 1973 δεν είναι η ίδια με τη 1975 για την ακτή του ελεφαντοστού ή για τις διάφορες άλλες που αφορούν το καγκό. Αυτό δείχνει ότι τον κύριο λόγο τον έχει η πολιτική. Ακόμη και το ΝΑΤΟ σε αυτήν υποτάσσεται. Ζητάνε η πολιτική από τον ΝΑΤΟ να εφαρμόσει την απόφαση. Το παράδειγμα της UFOR στη Λιβύη δηλαδή δείχνει ότι οι πολιτικοί δέχονται να παίξουν το ρόλο αυτό, να σταματήσει δηλαδή να υπάρξουν όρια στη στρατιωτική δράση κτλ. Things Δεν είναι αλήθεια ότι οι ανθρωπιστικοί δεν θέλουν καμία στρατιωτική παρέμβαση. Ο στρατηγός Γκανέσα μας το είπε ρητά ότι μπορούν να συνεννοηθούν οι δύο πλευρές. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν οι μένα να συνομιλήσουν με τους δε. Σε προβλήματα όπως της ΑΕΤΙΣ βλέπουμε ότι οι ανθρωπιστικοί μπορούν να ζητήσουν στρατιωτικούς πόρους γιατί στην περίπτωση εκείνη η στρατιωτική εκεί βοήθησαν την ανθρωπιστική δράση. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε να μην κάνουμε τέτοιου είδους γενικεύσεις. Δεν είναι ότι οι ανθρωπιστικοί δεν μιλάνε με τους στρατιωτικούς και το ανάποδο. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Έχουν κωδικοποιηθεί, οργανωθεί οι σχέσεις των δύο σκελών. και είναι ενδιαφέρον ότι το μάθημα που πήραμε από το Πακιστάν μέχρι τώρα ως προς το ΝΑΤΟ είναι ότι στο Πακιστάν το ΝΑΤΟ ήθελε να τα κάνει όλα εκείνο. Τους είπαμε προσέξτε γιατί υπάρχει σύγχυση. Η δική μας ευθύνη είναι να συνδυάζει τα δύο ως συντονιστής χωρίς όμως να παραβιάσει καμία από τις αρχές. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πλήρης κατανόηση των αρχών και η πολιτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική πλευρά θα καταλάβουν η μία τον ρόλο της άλλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρέμι έχει το λόγο που είναι εκτελεστική διευθύντρια της Oxfam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με καλέσατε, με προσκαλέσατε σήμερα. Και έτσι έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για την Oxfam και να σας πω πώς βλέπουμε τα πράγματα. Η Oxfam η Oxfam Novib είναι μέλος μιας συνομοσπονδίας της Oxfam που απαρτίζεται από 14 ανεξάρτητες οργανώσεις και συνεργαζόμαστε περί τις 80 χώρες για ανθρωπιστική βοήθεια σε μακροχρόνια βάση και για την ανάπτυξη και εκστρατείες. Μας ενδιαφέρει κατά καταπολέμηση της αδικίας και της φτώχειας. Η προσέγγιση μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν υπάρχει χώρος για την φτώχεια, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πολλά προελέχθηκαν και είμαι η τελευταία ομιλήτρια κατά το οποίο καθιστά το έργο μου ακόμα πιο δύσκολο γιατί θα πρέπει να φέρω να εισαγάγω νέα στοιχεία κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί τα περισσότερα προελέχθησαν και τα δέχομαι βεβαίως όλα. Είναι γεγονός ότι για την Oxfam δεν θα πρέπει να υπάρχει στρατιωτικοποίηση και πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάτι τέτοιο υποσκάπτει την ε, ίδια την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και την αξιοπιστία της διεθνούς κοινότητας. Διότι, όπως αναφέρθηκε, αυτό που έχει σημασία είναι πώς μας βλέπουν Οι άλλοι πώς μας βλέπουν οι διάφορες κοινότητες. Είναι θέμα αντίληψης. Και βλέπουμε ότι η πορεία μας δεν είναι καθόλου καλή. Το Φεβρουάριο συντάξαμε μία έκθεση ως Oxfam μιλώντας για το, με τίτλο «Για ποιανού βοήθεια πρόκειται» και αυτό μας ενδιαφέρει είναι οι εξελίξεις. Θα ήθελα να σας κοιογραφήσω αυτές τις εξελίξεις. που σχετίζεται με αυτά που σας προείπα. Αν πούμε τον τομέα της έρευνας, βλέπουμε ότι το 25% της αναπτυξιακής βοήθειας στο σύνολό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Το 25% τα τελευταία χρόνια αφορούσε τρεις χώρες, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Και πιστεύω ότι ο κατάλογος αυτός δείχνει ότι οι πολιτικές πεπιθήσεις ήταν να καθοριστικό στοιχείο για την χορήγηση της βοήθειας. Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση ε, αφορά το Ιράκ. Το 2008, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρωταρχικά τα κράτη-μέλη έδωσαν 5 δις δολάρια βοήθεια στο Ιράκ και το 2009 αφού αποχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις, η βοήθεια μειώθηκε από 5 εκατομμύρια, από 5 δις μάλλον θα εννοεί η ομιλήτρια, σε 225 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι επιθυμητό, διότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή συνδέονται άμεσα με θέματα πολιτικής υφής και με τις ε, πολιτικές πεπιθήσεις των ε, πάντων. Πολλοί αναφέρθηκαν στο Αφγανιστάν και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα, γιατί η χώρα αυτή <laughs> μας δείχνει ότι η προσέγγιση που ε, ε, λήφθη υπόψη δημιούργησε πολύ αρνητική εντύπωση και αποτελέσματα. Η Oxfam είναι δραστήρια στο Αφγανιστάν, Αφγανιστάν από το 1982. Έχουμε συνεργαστεί με ε, τοπικούς φορείς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Εγώ μόλις επέστρεψα από το Αφγανιστάν και αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η ατζέντα σε σχέση με τη μετάβαση και το μεταβατικό καθεστώς ως προς τις στρατιωτικές δυνάμεις και τις αναπτυξιακές, καθώς και τις ανθρωπιστικές, αυτά είναι τα τρία στοιχεία που ορίζουν την διαδικασία, το μεταβατικό αυτό πλαίσιο. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη ανθρωπιστική βοήθεια επειδή τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ε, μια εντολή, η Oxfam δεν μπορεί να αναλάβει ε, κυρίαρχο ρόλο ή ανεξάρτητο ρόλο, κάτι το οποίο θα ήταν ε, καθοριστικό. Εξαιτίας της μετάβασης αυτής της όθησης προς ένα μεταβατικό καθεστώς φαίνεται ότι θα υπάρχουν και άλλες ε, στρατιωτικές ε, δράσεις. Στο Χέλμαν δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν πλέον πληροφορίες. Πρόκειται για μία μαύρη τρύπα. Δεν υπάρχει καμία πρόσβασιμότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να χορηγήσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Η, η πρόσβαση είναι πολύ περιορισμένη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα, μια ανεξάρτητη ανθρωπιστική εντολή έτσι ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μπορέσουν να συμμετάσχουν, να γίνουν διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε επίπεδο πολιτών. Για να συνοψίσω, δεν λέω ότι έχουμε αποτύχει ολοκληρωτικά, θα πρέπει να αντιλήσουμε από τα διδάγματά μας, τα διδάγματα αυτά, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχει στρατιωτική προσέγγιση του θέματος, έτσι ώστε να διανύμουν εκείνη η ανθρωπιστική βοήθεια για να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Θα πρέπει να γνωρίζουν με τι θέλουν οι πολίτες να... και να τους στηρίξουμε. Γιατί διαφορετικά το χάσμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο μεταξύ των πληθυσμών και της ε, διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Και είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει χάσμα όχι μόνο μεταξύ πληθυσμού και διεθνούς κοινότητας, υπάρχει ολένα και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και της διεθνούς κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι όταν μιλάμε για μακροχρόνιες ε, εξελίξεις, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αναγκαία στοιχεία για να έχουμε μια υγιή mm-hmm. εξέλιξη. Εστιάσαμε όμως την προσοχή μας στη, στα βραχυπρόθεσμα ωφέλη. Τι βλέπουν ε, οι άνθρωποι επί που βλέπουν ότι ε, υπάρχουν δισεκατομμύρια βοήθειας που εισραίουν, αλλά δεν βλέπουν καμία βελτίωση στη χώρα τους. Άρα δεν φτάνουμε ούτε στους ε, πολιτικούς στόχους. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει τίποτα τα τελευταία δέκα χρόνια έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση του κύρους της ε, κυβέρνησης. Ούτε καν συμβαίνει αυτό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, έχει μεγάλη σημασία να χορηγείται βοήθεια ανεξάρτητα από άλλους φορείς και επίσης ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός μας θα πρέπει να είναι στοχοθετημένος, δηλαδή να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και να μείνουμε μακριά από την πολιτική ατζέντα. Δεν μπορούμε να υπαγάγουμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε πολιτικούς στόχους ή ιδεώδη. Για μένα αυτό είναι απόλυτα σαφές. Ελπίζω η ΕΚΟ να το συνειδητοποιήσει και να παραμείνει ανεξάρτητη. Τέλος, ε, ως προς το στρατιωτικό σκέλος, τη U4, θα πρέπει να επέμβει μόνο εάν είναι απολύτως αναγκαίο. Θα πρέπει να μην υπάρχει καθαρά στρατιωτική παρέμβαση όπως βλέπουμε τώρα και στη Λιβύη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρέντς ή Γκέρεντς Οι τρεις αυτές παρεμβάσεις δεν μας διευκολύνουν τα πράγματα. Επανέρχομαι λοιπόν στα ερωτήματα που έθεσα πριν. Δικαίως λέτε ότι σε μερικές περιπτώσεις οι στρατιωτική και οι ανθρωπιστική συνεργάζονται πολύ καλά, όπως στην ΑΕΤ. Αυτή η περίπτωση όμως διαφέρει πολύ από την περίπτωση μιας σύραξης που μπορεί να συμβεί αλλού. Το αντίθετο μάλλον, δεν συνεργάστηκαν καλά. Σε άλλες περιπτώσεις σύραξης όμως, χωρίς τους στρατιωτικούς δεν θα γινόταν τίποτα. Και όποια ανθρωπιστική βοήθεια χορηγηθεί θα οφείλεται στους στρατιωτικούς. Από την άλλη, η κυρία Καρίμη, εσείς βλέπετε τα πράγματα με πολύ μεγαλύτερη φρόνηση από τους υπόλοιπους δύο. Θα ήθελα να μου πούν και οι τρεις το εξής. Στο ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει οτιδήποτε ώστε να μπορέσουν οι τρεις παράγοντες να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή μήπω το σύστημα που έχουμε δεν είναι το καλύτερο. Και προς τον εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν τόποι όπου και εσείς μπορεί να χρειαστεί να αποσυρθείτε παρά το ότι έχετε αυτόν τον αναγνωρισμένο ουδέτερο χαρακτήρα. Τι μπορεί να σας οθήσει να αποσυρθείτε από κάποιον τόπο. Πού βρίσκονται τα όρια που ούτε εσείς δεν μπορείτε να ξεπεράσετε. Ποιος θέλει να αρχίσει. Ορίστε εσείς κύριε Λακούρο. Ποια είναι τα όρια. Υπάρχουν περιπτώσεις πράγματι όπου δεν υπάρχει απλώς πρόσβαση για λόγους ασφαλείας στους πληθυσμούς που θα θέλαμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι σαφές. Τι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι συνηθισμένος να δράσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προσαρμόζονται σε δύσκολες συνθήκες σε καταστάσεις όπου η ασφάλεια δεν είναι άριστη. Η διαφορά όμως είναι ότι είναι μεταξύ του να καταστεί κανείς θύμα του περιβάλλοντος ή του να καταστεί θύμα επιθέσεων. Εδώ υπάρχει όριο. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες οργανώσεις. Όταν κανείς γίνεται θύμα άμεσων επιθέσεων σταματούν οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι σαφές. Στον γενικότερο ανθρωπιστικό χώρο η κοινότητα υπάρχουν διαφορετικές αντιστάσεις. Ο ΙΕ έχει ένα σύστημα ταξινόμησης του κινδύνου και εμείς όχι γιατί είμαστε πιο θαραλέοι αλλά γιατί είμαστε άλλη οργάνωση έχουμε άλλο και συνήθως παραμένουμε πιο πολύ καιρό επί τόπου. Σε τέτοιες καταστάσεις όπου χρειάζεται να αποσυρθούμε κάποτε θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία πολιτική προσέγγιση ως προς το ποια είναι τα όρια γι' αυτό φεύγουμε όταν δεν μπορούμε πια να επιζήσουμε σε τέτοιο περιβάλλον. Ξέρω ότι ορισμένοι παράγοντες, για ορισμένους παράγοντες, το ότι είμαστε ουδέτεροι, ανεξάρτητοι και αυτά όλα τα αποδεικνύουμε από τη δράση μας και ότι είμαστε και αδέκαστοι, μας μας καθιστά προτιμητέους. Εγώ δεν ανήκω βέβαια σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, αλλά συνεργάζομαι με αυτά. Το ερώτημά σας λοιπόν ήταν αν ε, είναι κατάλληλο το περιβάλλον, το νομικό, νομοθετικό περιβάλλον που υπάρχει στην Ένωση ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διεκπαιρέωση των καθηκόντων μας. Ε, όπως είπε και ο Πέτρος Σανκόρ το πρωί, νομίζω ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όσοι έχουν σήμερα και με τις δικαιοδοσίες της κυρίας Επιτρόπου για τα ανθρωπιστικά δείχνουν ότι η εξωτερική υπηρεσία δεν κάνει τα ίδια με την Κομισιόν ούτε το Κομισιόν με το Συμβούλιο. Και στην Ολομένεια στις 18 Ιανουαρίου και εσείς υπενθυμίσατε ποιες είναι οι ανθρωπιστικές αλλά και πολιτικές σας υποχρεώσεις. Έχετε νομίζω κατάλληλα, τα κατάλληλα εργαλεία αλλά υπάρχει και θέμα συγκυρίας. Άλλο η Αιτή, άλλο η Λιβύη και άλλο το Τσάντ. Επίσης σημαντικό είναι να μας οδηγούν μένει οι αρχές αυτές αλλά να είμαστε και σε θέση να δηλώσουμε, να παρεγράψουμε ότι στο α περιβάλλον δρούμε με τρόπο α και στο β με β γιατί μερικοί λένε γιατί δέχεστε τους στρατιωτικούς στην ΑΕΤ και τους καλείτε και μόνοι σας και στη Λιβύη δεν τους θέλετε. Δεν είναι θεσμικό μόνο αυτό το πρόβλημα, αν και νομίζω ότι φάνηκε από την ΑΕΤ ότι αποσαφηνίζεται ο ρόλος του Monitoring Information Center και των υπολείπων παραγόντων. Νομίζω ότι είναι θέμα διαλόγου και αμοιβαίας συνεννόησης και κατανόησης. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα μερικοί πρεσβευτές στο ΚΟΠΣ που λένε ότι το πράγμα έχει ξεπεράσει τα όρια. Ότι δηλαδή το ότι είμαστε ένας δείκτης των αποφάσεων του ΚΟΠΣ για το κατά πόσον θα δράσουν οι στρατιωτικοί αποσιοποιητικά. Υπάρχει όμως και άλλο θέμα, μπορεί να χρειάζεται και άλλη προσπάθεια ώστε τα θεσμικά όργανα να καταλάβουν ότι εδώ πρόκειται για συνεργασία πολλών παραγόντων. Δεν μπορείτε να μας πείτε ονόματα. Η κυρία Καρυμή. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είπα απλώ ότι από το 82 είναι η Oxfam στο Αφγανιστάν. Δηλαδή είμαστε εκεί πολύ πιο πριν από τους ε, στρατιωτικούς και θα είμαστε εκεί και μετά το 2014. Εγώ πήγα πρώτη φορά το 2000 στο Αφγανιστάν. Και υπό τη διοίκηση των Ταλιμπάν τότε. Από τότε πήγαινα τακτικά. Διαπίστωσα δε ότι δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό το πρόβλημα εκεί έχουμε και πολιτικά προβλήματα, θέματα πολιτικής ατζέντα. Δεν μιλάμε μόνο για διαφοροποίηση μεταξύ ατζέντα ανθρωπιστικής και πολιτικής, πράγμα απαραίτητο να γίνει, αλλά πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να επιτύχουμε μέσα από τις δράσεις μας σε αυτές τις καταστάσεις. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι πολύ πιο μετριοπαθής Δηλαδή μην νομίζει ότι μπορεί να επιφέρει και τεράστιες αλλαγές μέσα από στρατιωτική δράση, δεν συμβαίνει αυτό, πάντα αυτό. Ε, εκτός αυτού μιλήσατε και για το θεσμικό σύστημα. Αυτό που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι γραμμές του προϋπολογισμού Πού χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Υπάρχει ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός βέβαια που είναι αρκετά σημαντικός, αλλά εδώ καταπολεμούμε τη φτώχεια και ο βασικός στόχος δεν είναι να προβάλλουμε τους πολιτικούς στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι με όλη αυτή τη συζήτηση για τη θέση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την κατάταξή της, το ρόλο της, πρέπει να φροντίσουμε να μην υποταχθεί στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης η ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική. Αυτό θα ήταν πολύ επιζήμιο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος των εργασιών μας. Euh, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, προσκαλεσμένους μας, όλους τους ομιλητές όλους όσους συμμετείχαν. Χαίρομαι γιατί τα καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση με ανταλλαγή απόψεων και βλέπουμε ότι εξελίσσονται τα πράγματα προς το καλύτερο ως προς τη συνεργασία στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους Και θα ήθελα να πω, όπως είπε και ο στρατηγός, ε, τηρούμε και πιστεύουμε οι μεν στους δε. Έχει σημασία, πολύ μεγάλη σημασία η ουδετερότητα των πηγών χρηματοδότησης, έτσι δεν είναι κύριε Γκέρενς, ε, αλλά επίσης να γνωρίζουμε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, και, ουδέτεροι και αμερόληπτοι, ό,τι και να συμβαίνει. Σας εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την εργασία και να ξαναβρεθούμε σε μια μελλοντική ακρόαση, ε. γιατί προχωρήσαμε αρκετά και γι' αυτό θα χρειαστούν και άλλες ακροάσεις για να δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.